Αν ήρθαν τα μέλη μπορούν και να καθίσουν. παρακαλώ να καθίσετε και να λάβετε θέσεις. Δεν θα κάνω τις ανακοινώσεις του Προέδρου όσο μιλάτε μεταξύ σας. Thank you very much. This is a continuation of our meeting. Συνεχίζουμε την χθεσινή μας συνεδρίαση και γι' αυτό ως ήθιστε θα κάνω τις σοβαρές ανακοινώσεις από την αρχή οπότε και θα είναι οι βουλευτές παρόντες. Ορισμός μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Σώματος για τη Στατιστική. Στατιστική. Οχτώ από τους δώδεκα ζητούν να γνωμοδοτήσουμε για τον ορισμό τους. γιατί η Επιτροπή, αυτή η Συμβουλευτική Επιτροπή λίγη θητεία της σε λίγο. Έχουν προεπιλογή 8 από τους υποψηφίους από τους συντονιστές της εικόν και των Λίων Γκόκ. Αλλά δεν ξέφρασαν καμία αντίρρηση στα προτινόμενα ονόματα. Βιογραφικά τους έχουν διανεμηθεί σε όλους. Εκτός εάν λοιπόν δηλώσετε την αντίρρησή σας θα θεωρήσουμε ότι ότι θα εγκρίνονται και θα στείλω επιστολή στον πρόεδρο λέγοντας ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα, οι συνεχιζόμενοι τριμερείς διάλογοι. Μα πάλι μιλάτε. Γιατί μιλάτε. Αν θέλετε να ψηφίσουμε πρέπει να σταματήσετε τις συνομιλίες. Λοιπόν, δεύτερος τριμερής διάλογος 4 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο και εξέτασε τα παραμένοντα εκκρεμή θέματα που αφορούν κυρώσεις και μισθούς. Για το AIFMD ιδίω. Παρακαλώ, αν θέλετε να συνομιλείτε θα σταματήσω εγώ, να το ξέρετε. Είπε λοιπόν το Συμβούλιο ότι και για το MIFID και για το AIFMD και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να τα ξανασκεφτούν και να καταλήξουν στις 26 Φεβρουαρίου εν Εστρασβούργο. Όταν σταματήσετε να συνομιλείτε τότε θα συνεχίσω. Ορίστε μας. Εγώ κάνω τις ανακοινώσεις της Προέδρου και δεν, συνο... στατιστική για τα διάφορα επαγγέλματα intertrained. Έγινε και αυτό ο τριμερής διάλογος και καταλήξανε σε συμφωνία με το Συμβούλιο για τα περισσότερα θέματα εκτός από την επιτροπολογία διότι το Συμβούλιο θέλει να αλλάξει τα πράγματα ενώ το, ε, το Κοινοβούλιο θέλει κατεξουσιοδότηση πράξη. Για τον ανταγωνισμό η πρώτος τριμερής διάλογος συζήτησε τις αποζημιώσεις για παραβιάσεις ανταγωνιστικό νόμο ή στον νόμο για την ανταγωνιστικότητα και για τη σύνδεση μεταξύ αποζημιώσεων και προστήμων. Και στις 27 Φεβρουαρίου θα συνεχίσει ο διάλογος αυτός, ελπίζουμε να, τότε να καταλήξουμε. Μέχρι τώρα τα πράγματα πήγαιναν πολύ καλά από, από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Ήταν ο πρώτος τριμερής διάλογος και συναπόφαση για τον ανταγωνισμό. Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία για τις στατιστικές, για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, το σημείο 11 δηλαδή. Αν φέρατε τις κάρτες σας μπορείτε και να ψηφίσετε. Για να κάνουμε μια πειραματική ψηφοφορία, δοκιμαστική. Είχατε θέσει το θέμα του τριμερούς διαλόγου usage και μόλις διάβασα στους Financial Times κάτι, το Συμβούλιο δεν ζητάει ευθυγράμμιση των κυρώσεων μόνο με το MIFID, αλλά επιλεκτικά οποτεδήποτε εφαρμόζεται το χαμηλότερο δυνατό πρότυπο. Αλλά δεν συμφώνησαν όλοι, ιδίως στην ομάδα μου και το θέτω διότι δημιουργεί μερικές ανησυχίες στον τύπο γιατί δεν καταλήγει η συζήτηση. Δεν καταλήγει γιατί το Συμβούλιο δεν θέλει τα ίδια πρότυπα κυρώσεων που θέλουμε και εμείς. Και εμείς δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε αυτά όλα ταυτόχρονα όσα έχουμε συζητήσει, να το ξέρετε αυτό. Είμαι ανοιχτό σε συμβιβασμούς, αλλά Γι' αυτό πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις και οι δύο πλευρές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δοκιμαστική ψηφοφορία. cards plugged in that are not responding. Δύο κάρτες φαίνεται δεν δουλεύουν. Λοιπόν. Yeah. That's that closed right. Clear that. So, first of all, um... Λοιπόν, τώρα τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική γ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική δ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση επαλήθευση απορρίπτεται Συμβιβαστική σιγματάφ F υπέρ. Συμβιβαστική σιγματάφ F υπέρ. Κατά. Ποιες εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίζουν περισσότεροι, αλλιώς δεν βλέπω καλά τι γίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Α, δεν βλέπω, δεν βλέπω. Λοιπόν, επαλήθευση ηλεκτρονικά. Και παρακαλώ να πάψουν οι ιδιωτικές συζητήσεις. 26. θα προσθέσουμε μία ψήφο υπέρ. Λοιπόν, έληξε, εγκρίνεται σχεδόν ομόφωνα 87 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 27 έχει αποσυρθεί απασχόλησης 10 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική ζήτα G υπέρ. Κατά. Χες. Ήτα υπέρ. Κατά. Αχ Παναγία μου. Επαλήθευση. Γιατί δεν βλέπω χέρια. Αν ψηφίζετε και για άλλους, Μα είπα συμβιβαστική ήταν, γιατί δεν έβλεπα τα χέρια. Άλλοι τρεις ακόμα, άντε, έληξε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Ι Ι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική J, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Κ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περίφ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβ, συμβ, α, επαλήθευση, καλά, επαλήθευση για την 33. Ένας ακόμα κατά, εντάξει, απορρίπτεται. Συμβιβαστική λάμδα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περίφ 3 υπέρ, Θα συνεχίσω όταν σταματήσετε είπα. Περίφ 3 υπέρ κατά αποχές α δεν κατάλαβα επαλήθευση για την περίφτρια περίφτρια παύλα 3 α νέα εγκρίνεται συγγνώμη πολύ δύσκολη αίθουσα εδώ για να βλέπει ο πρόεδρος. Και γιατί συζητάτε μεταξύ σας βρε παιδιά. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, επαλήθευση, επαλήθευση. Επαλήθευση. «23 με 15 εγκρίνεται. Περίφ 4 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση εγκρίνεται χιχι συμβιβαστική μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επαλήθευση για την νη. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική όμικρον υπέρ. Συμβιβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περίφ 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική ρο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απασχολήσεως 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παλήθευση άμα θέλετε εντάξει. Παλήθευση. Αν ένας ακόμα Έληξε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 32 με 5. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Περίφευτα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται περίφ 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται περίφε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται περίφ 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά άποχες επαλήθευσης Έληξε. Εγκρίνεται. 13, περίπου 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 14 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίν, απορρίπτεται, 32 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικά το σύνολο όπως τροποποιήθηκε. ...38 υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή για το νομοθετικό ψήφισμα. ψήφος ακόμα ένας, 36 υπέρ, μία ψήφος κατά καμία αποχή. Το Μάρτιο στην Ολομέλεια. Ε, πάμε λοιπόν τώρα στην έκθεση Giggold. Θα αλλάξουν οι υπάλληλοι εδώ, τι θα γίνει. Α, ναι. Καλώς, είναι όλοι έτοιμοι. Συμβιβαστική AC σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα του AC ψηφίσατε όλοι δεκτή τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. AD ε, τώρα η συμβιβαστική στη σελίδα 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Πηγαίνουμε τώρα στην 168 Πρώτο τμήμα υπέρ. Για μια στιγμή. Λοιπόν, 168 ως έχει, ψηφίζουμε. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 168. Amendment 168 and others. Voted, Ψηφίσατε όλοι, τέλος. Δεκτή. Οι υπόλοιπε καταπίπτουν, αλλά να δω μέχρι πού. Πηγαίνουμε τώρα στο AE, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτό. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το πέμπτο τμήμα της AE. Voted and that's carried. Δεκτή έκτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έβδομο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Θέλετε να υπάρξει έλεγχος. Κοιτάξτε, κανονικά πρέπει να δείχνετε με τα χέρια σας τι θέλετε να κάνετε. Πέρα τη ψηφοφορίας δεκτό. Για το 8ο τμήμα. Σηκώστε τα χέρια σας να βλέπω λέει πρόεδρος. 8 υπέρ. Βέρνερ δεν έρχεσαι να προεδρεύσεις καλύτερα. Ζων Πολ πες του πόσο εύκολο είναι να βλέπει κανεί την ψηφοφορία πώ πηγαίνει σε μια τέτοια αίθουσα. Θέλετε να τα αναβάλουμε για την επόμενη εβδομάδα για καλύτερη αίθουσα, τι ναι. θέλετε. Λοιπόν, οκτώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 8ο τμήμα της AE. Πέρας της ψηφοφορίας. Καταπι... Ε, μάλλον απορρίπτεται. Ένα το τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το ένα το τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτή. Πηγαίνουμε τώρα στην 185. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική AF. Με μία προφορική εδώ τροπολογία. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ποιοι είναι υπέρ. σε πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ευχαριστώ. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Δεκτό. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 212. Ποιοι είναι υπέρ της 212. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γιατί 212 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε όλοι. Τέλος. Δεκτή. Χωρίς μικρόφωνο σχόλια. Σας έδωσα όλες τις ευκαιρίες, λέει η Πρόεδρος. Τα είπα όλα αυτά πριν από εσά. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να ελέγξω εκ νέου. Συμβιβαστική AG σε διάφορα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πηγαίνουμε τώρα στο AH, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές δεκτή, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές δεκτό. Τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το τέταρτο τμήμα της AH. H. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίφθηκε. Πέμπτο τμήμα υπέρ. κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το πέμπτο τμήμα. Γίνονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα εδώ. Απορρίπτεται. στο AI υπέρ κατά αποχές δεκτή Περιμένω τους Γερμανούς να τελειώσουν τις συζητήσεις τους, λέει η Πρόεδρος. Ε, Τελειώσατε παρακαλώ. Συμβιβαστική AJ, τώρα σε τρία τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό, δεύτερο τμήμα υπέρ, <clears throat> κατά, αποχές, δεκτό, τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Πηγαίνουμε τώρα στην 122. Ποιοι είναι υπέρ, Α, όχι, έχει καταπέσει μου λένε εδώ. 3.34 υπέρ. Τροπολογία 3.34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Δεν ξέρω τι έκαναν βέβαια οι σοσιαλιστές, δεν είδα τα χέρια τους. Ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την 334. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απερίφθη. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Το αρχικό κείμενο παράγραφος 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξω ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. Γίνεται δεκτή 18 υπέρ 17 κατά. Το αρχικό κείμενο στην παράγραφο 4 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό αιτιολογικές σκέψεις ομαδών 1 με 20 υπέρ, κατά, δεκτές, τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, ομαδικά από 21 με 24 υπέρ, κατά, αποχές δεκτές, τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 2, Απερίφθη, συγγνώμη, λάθος. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 3. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 4. Ναι. Συμφιβαστική Α, πρώτο τμήμα. Carried part Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική C υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ή e πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω τι κάνει το ΕΛΚ, πρέπει να προβούμε σε ηλεκτρονική επαλήθευση. Είμαστε στο δεύτερο τμήμα της ε, συμβιβαστικής Ή, e, παρακαλώ. Ε. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η παρακαλω ψηφισατε ολοι Εγκρίνεται. Η συμβαστική GH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 326 υπέρ κατά αποχές ε, δυστυχώς πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 326. 326. Απορρίπτεται. Η 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβαστική J. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Εγκρίνεται. Πάμε στη 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική KL προφορική τροπολογία θέλετε να την παρουσιάσετε με την προφορική τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στη συμβιβαστική M. Υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβιβαστική NO. Υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβιβαστική PQ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στη συμβιβαστική RS. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές ε, ηλεκτρονική παλήτευση για το δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στη συμβιβαστική TX, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής TX παρακαλώ. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική Y Πρώτο τμήμα με προφορική τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην συμβιβαστική ZAB. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του κειμένου ως τροποποιήθηκε. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Εγκρίνεται. 33 υπέρ, 4 κατά, καμία εποχή. Πολύ καλή δουλειά, Σβέν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδης ηγητές και να πω χαίρομαι πάρα πολύ που οι περισσότεροι τάσσονται για μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή εποπτεία και αυτό επιβεβαιώθηκε φυσικά με τη βοήθεια όλων σας. Ο Σαρών, έχω μία ερώτηση επί διαδικαστικού. Δηλαδή, στην ΕΚΟΝ, στη δική μας Επιτροπή, ε, πότε θα μιλήσουμε για μία υποεπιτροπή. Γιατί τον Ιανουάριο είπαμε ότι είναι πλήρης επιτροπή και δεν νομίζω ότι ε, το Προεδρείο μπορεί να αποφασίσει με βάση μια επιστολή που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ το θέμα αυτό να τεθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης φοράς. Νομίζω, λέει η Πρόεδρος, ε, ζήτησα τους συντονιστές να το σχολιάσουν και το συζητήσαμε, νομίζω το συζητήσαμε. Όχι, λέει ο κύριος Λάγκε. Εντάξει, αν ε, θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να βάλω το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Αλλά όχι τώρα, για άλλη φορά αν θέλετε να καταψηφίσετε και να διαφωνήσετε με τη θέληση της διάσκεψης των Προέδρων, παρακαλώ. Δεν έχω καμία αντίρρηση, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Λάγκεν. Κοίτα, το μικρόφωνο παρακαλώ. Κοιτάξτε, η σύσταση μίας επιτροπής ε, είναι προνομία της Ολομέλειας και τον Ιανουάριο αποφασίσαμε ότι η Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, θα παραμείνει. Δεν θα γίνει υποεπιτροπή. Η υποεπιτροπή μπορεί να προταθεί από την Ολομέλεια στο Προεδρείο μόνο αν υπάρχει η ψηφοφορία της αρμόδιας επιτροπής. Άρα δηλαδή ε, δεν υπάρχει βάση για την απόφαση των προέδρων των πολιτικών ομάδων γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν ψηφίσει επ' αυτού και παρακαλώ να τηρήσουμε τη διαδικασία. Το Προεδρείο μπορεί να ψηφίσει μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η δική μας η ψηφοφορία και παρακαλώ το θέμα να αναβληθεί μέχρι να έχει ψηφίσει η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Πρόεδρος, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή τη φάση Λόγω της ε, ψηφοφορίας ε, στην Ολομέλεια που έλαβε χώρα στο πλαίσιο μιας έκθεσης ε, της Επιτροπής ΑΦΚΟ του να συσταθεί δηλαδή υπό Υποπιτροπή η διάσκεψη των Πρόεδρων μου ζήτησε για τρίτη φορά να καταθέσω κάποιες προτάσεις εφόσον έχουν απορριφθεί οι δύο προηγούμενες που είχαν κατατεθεί και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Επιτροπή αυτή δεν θέλει να αλλάξει. Εμείς λοιπόν ε, καταθέσαμε στη διάσκεψη των Προέδρων μία πρόταση για διαβουλεύσεις και εκείνοι κατέληξαν, είχαν πει ότι θα καταλήξουν ε, σε ένα συμπέρασμα, αλλά δεν κατέληξαν από αυτού και όταν καταλήξουν θα έρθει εδώ η πρότασή τους. Αυτή δηλαδή είναι η διαδικασία. Αυτοί μας ζητούν να καταθέτουμε προτάσεις, ε, να μας επιβάλλουν κάτι και Ό,τι και αν διαβάσει κανεί τον τύπο για προτάσεις της Bowles, κατ' ουσίαν είναι προτάσεις ε, τις οποίες ε, έχει ε, προετοιμάσει η Γραμματεία και έχουν εγκρίνει οι συντονιστές. Γιατί τέτοιου είδους διαδικασίες γίνονται συνεχώς. Δεν πρόκειται για τετελεσμένο γεγονός και σε κάθε φάση η προτίμηση να μην υπάρξει καμία αλλαγή, προφανώς και είναι η βούληση αυτής της Επιτροπής και εμείς το επιβεβαιώνουμε αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εγώ τουλάχιστον έτσι την ερμηνεύω. Αν τώρα εσείς ε, θέλετε συζήτηση από αυτού, πάρα πολύ ωραία και μπορούμε αν θέλετε να κάνουμε μια ενδεικτική ψηφοφορία και να ενημερώσουμε τη διάσκεψη των Πρόεδρων. Αλλά όλη αυτή η φασαρία και το μπέρδεμα προκλήθηκε λόγω της ψηφοφορίας στην Επιτροπή ΑΦΚΟ. Ούντο, έχει το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ Σάρων. Εγώ ε, βεβαίως ε, και είμαι πρόθυμος ε, να κρίνω όλους τους προέδρους πρωί και βράδυ, αλλά όταν ασκώ κριτική ε, θέλω να έχω κάποια στοιχεία στα χέρια μου. Και αυτή τη στιγμή θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν είμαι συντονιστής, όμως εδώ στην αίθουσα υπάρχουν αρκετοί συντονιστές. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα, από ό,τι κατάλαβα από τη συζήτηση, Αυτά που είπε η Σάρον με την ιδιότητά της της Πρόεδρου, Ακριβώς αυτά αποφάσισαν και οι συντονιστές στην Επιτροπή μας. Βέρνερ, εσύ δεν είσαι συντονιστής. Εάν λοιπόν αυτά δεν ισχύουν, τότε θα πρέπει να μας ενημερώσουν οι ε, συντονιστές. Ε, γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ αυτή τη στιγμή μην ε, επιδεικνύεται ιστερική στάση, νυφάλιοι να είσαστε. Η Σάρον έκανε αυτά που αποφάσισαν οι συντονιστές. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν για αναταραχή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ε, επανεξετάσουμε το θέμα. Αλλά καταρχήν ας παραμείνουμε όπως σας είπα νυφάλιοι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι όποιος είναι λογικός και αυτό ισχύει ως βασική προϋπόθεση. Όποιος είναι λογικός Κανείς δεν μπορεί να πει στην Επιτροπή αυτή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να ασχολείται με την Ευρωζώνη και με τις διάφορες ενδιάμεσες λύσεις που εξευρίσκονται. Δηλαδή, δεν θέλετε να έχετε καθόλου λέγει στο πώς ε, θα χαράσουν τα κράτη-μέλη την πολιτική τους στην Ευρωζώνη. Αν ε, θέλετε να βρείτε μία θεσμική απάντηση, Βεβαίω το ποια είναι η σωστή απάντηση, επ' αυτού να, μπορούμε να συζητήσουμε και εγώ δεν έχω αποφασίσει επ' αυτού. Η συζήτηση όμως να γίνει επί της ουσίας και όχι μέσα από αυτή την αναταραχή, γιατί νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα βοηθήσει κανένα. Βέρνερ, εσύ ήδη πήρες το λόγο και τώρα έχουν στήσει το λόγο άλλοι. Ο Ότμαρ έχει στήσει το λόγο και μετά ο Σβέν. Θα συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο κύριος Μπούλμαν. Υπάρχουν ε, τρία επίπεδα και εγώ θα προσθέσω και ένα τέταρτο. Δηλαδή, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι αποφάσισαν οι συντονιστές. Μόνο που αν έχουν αποφασίσει κάτι, τότε αυτό αντίκειται σε αυτό που είπε τώρα μόλις η πρόεδρος, ότι δηλαδή η πλειοψηφία της Επιτροπής μας είναι κατά μιας ε, υποεπιτροπής. Θα ήθελα όμως ε, να γνωρίζω πώς ακριβώς έγινε η συζήτηση ανάμεσα ε, στην πρόεδρο και τους συντονιστές. Εγώ δεν θεωρώ ότι η πρόεδρος έδρασε με δική της πρωτοβουλία τη στιγμή μάλιστα που γνωρίζει ότι η Επιτροπή έχει διαφορετική άποψη. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Εφόσον υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας η διάσκεψη των Προέδρων ε, δεν μπορεί να γνωρίσει την απόφαση της Ολομέλειας και έτσι φτάνουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο. Όχι μόνο στη σχέση της Επιτροπής προς τη διάσκεψη των Προέδρων αλλά και προς τη σχέση της διάσκεψης των Προέδρων προς απόφαση της ε, Ολομέλειας. Βεβαίως ε, μπορούμε να κάνουμε έτοιμα προς την Ολομέλεια να αναθεωρήσει την απόφασή της, αλλά δεν υπάρχει κανένα όργανο που να μπορεί να ανακαλέσει απόφαση της Ολομέλειας. Και το τρίτο θέμα που έθιξε ο κύριος Μπούλμαν αφορά στη νόμιμοποίηση, ε, στο να μπορούμε να εκφράσουμε άποψη σε θέματα Ευρωζώνης. Νομίζω μέχρι τώρα έχουμε πει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα συμβάλλει στην διάσπαση της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ευρωζώνη και εκτός Ευρωζώνης. Εμείς ε, θεωρούμε ότι αυτό το Κοινοβούλιο ενώνει και δεν διασπά την Ευρώπη. Για μένα μέχρι τώρα Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το Κοινοβούλιο ήθελε να έχει λέγην για όλα τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό επιμένει το Κοινοβούλιο να εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο. Θα συνεχίσουμε με τη συγκεκριμένη υπόθεση γιατί δεν θα περάσουμε στη συζήτηση κανονικά αυτή παρά την επόμενη ώρα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι συνεισφορές σας θα πρέπει να βασίζονται στο έγγραφο και όχι σε κάποιες αναφορές. για διάφορα τα οποία αφορούν αποκλειστικά την Ευρωζώνη. Σβέν. Νομίζω ότι υπάρχουν εδώ δύο επίπεδα ε, ενεργειών από τη μία αυτά που έχουν κάνει οι συντονιστές και από την άλλη επί της ουσίας. Για τους συντονιστές υπήρξαν δύο διαφορετικές παρεμβάσεις. Αν κατάλαβα καλά τη συζήτηση στους συντονιστές υπήρξε μια αρκετά σημαντική συμφωνία ότι στο μέλλον μπορεί να χρειαστούμε μια υποεπιτροπή. Το θέμα είναι αν ε, εμείς σαν κοινοβούλιο θα πάρουμε την απόφαση που θα δεσμεύει το επόμενο κοινοβούλιο και εμείς εξεπλάγημε σαν πράσινοι στη διάσκεψη των Προέδρων που αποφάσισε το πώς θα οργανωθεί το επόμενο κοινοβούλιο. Η επιστολή σας, Πρόεδρε, δεν έλεγε να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Και γι' αυτό ο Γενικός Γραμματέας μας ζήτησε να αναβληθεί η ψηφοφορία. Αυτό έγινε και ανοίγει την δυνατότητα για μια καλή συζήτηση. Πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση και με τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος γιατί είναι θέμα που αφορά το σύνολο της Επιτροπής και όχι μόνο τους συντονιστές. Αυτά για το διαδικαστικό. Επί της ουσίας τώρα. Πράγματι, ε, σε σχέση με τον έλεγχο του Eurogroup, εμείς έχουμε πολύ λίγα δικαιώματα. Έχουμε στην ουσία μια de facto ε, ευρωζωνική κυβέρνηση, θα έλεγα, η οποία δεν ελέγχεται από κανένα δημοκρατικά. Το θέμα είναι θα δημιουργήσουμε νέες δομές ενώ δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Η έκθεση της Τρόικας ζητά να εφαρμοστούν τα κοινοβουλευτικά δικαιώματα. Εμείς επανειλημμένα καλούμε υπουργού εδώ οι οποίοι και αν έλθουν όταν έρχονται δεν μας δίνουν τις απαντήσεις τους. Λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουμε τι περιθώριο κίνησης έχουμε ε, στα πλαίσια των νομικών δεσμεύσεων. Ξέρουμε ότι πράγματι για νομικούς λόγους δεν μπορούμε να διακρίνουμε εμείς τα μέλη της Ευρωζώνης από τα υπόλοιπα μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε την κατάσταση, να σεβαστούμε τις διάφορες χώρες, αλλά ταυτόχρονα να σεβαστούμε και τα κοινοβουλευτικό μας δικαιώματα και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ένα ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης, Πρόεδρε. Όχι μόνο η επιστολή σας, αλλά μια γενικά συζήτηση για τα δημοκρατικά δικαιώματα του Κοινοβουλίου να ελέγχει το τι συμβαίνει και στην Ευρωζώνη. Ο Ζων Πολ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν αυτά που είπε ο Σβέν συμφωνούν με αυτά που συζητήθηκαν στους συντονιστές. Θα ήθελα να σας πω ακριβώς τι υπόθηκε. Καταρχήν, ότι η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να τα δει σφαιρικά τα πράγματα και να μην τα διαιρέσει. Δεύτερον, ότι δεν ήταν, θα ήταν σωστό να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα να προταθούν πριν λήξει η θητεία. Και τρίτον, ότι η δυνατότητα δημιουργίας μιας υποεπιτροπής συζητήθηκε μεν ως μία πιθανή λύση, με βάση όμως δύο νομικά θέματα. Ένα, η υποεπιτροπή αυτή δεν μπορεί να ιδρυθεί παρά με την πρωτοβουλία της προϋπάρχουσας επιτροπής στο επόμενο κοινοβούλιο, άρα δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε σήμερα να, αποφα... να ιδρύσουμε υποεπιτροπή. Και δεύτερον, για τους λόγους που ανέφερε ο Σφεν και ο Ότμαρ, οι βουλευτές εκπροσωπούν το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών και δεν υπάρχει καμία νομική βάση για να τους διαχωρίσουμε με βάση τη ζώνη όπου εκλέχθηκαν, αν εκλέχθηκαν μέσα ή έξω από την Ευρωζώνη δηλαδή. Αυτά είναι οι βάσεις του συστήματος. Τώρα, δεν μπορούμε παρόλα αυτά να γνωρίσουμε ότι υπάρχει ένα αίτημα να γίνει έλεγχος για τα απεπραγμένα της Ευρωζώνης και εκτός αν δημιουργηθεί δεύτερο κοινοβούλιο μόνο για την Ευρωζώνη ο μόνος τρόπος θα ήταν ο δρόμος που αφήσαμε ανοιχτό, δηλαδή μία συμφωνία κυρίων που να μία συμφωνία κυρίων λοιπόν που αν δημιουργηθεί αυτή η υποεπιτροπή να δίνει προτεραιότητα στους βουλευτές της Ευρωζώνης χωρίς να αποκλείονται οι υπόλοιποι. Απαιτείται λοιπόν ε, μία προσπάθεια συμβιβασμού και συμφιλίωσης εδώ. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Ούτως ή άλλως η δημιουργία υποεπιτροπής δεν μπορεί παρά να ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή του επόμενου Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Επόμενο. Πολύ σύντομα συμφωνώ με αυτά που είπαν ο Σβέν και ο Ζαν Πολ. Έχουμε ένα νομικό πλαίσιο γνωστό, εγνωσμένο. Πρέπει να το σεβαστούμε, αλλά συμφωνώ με τον Σβέν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα λογοδοσίας και ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε αυτά που υπάρχουν. Αν δεν δείξουμε ένα βαθμό ευελιξίας, τότε θα δημιουργούνται συνεχώς, θα παίρνονται αποφάσεις εκτός ημών ενώ στα τραπεζικά θέματα είμαστε σε συναπόφαση. Προσπαθήσαμε ως συντονιστές να υπενθυμίσουμε πώς έχει το δίκαιο και θα αποφασιστεί ό,τι αποφασιστεί συλλογικά, όχι ένας. Δεν θα αποφασίσει ένας. Γιατί μπροστά μας έχουμε ίσως την πιο δύσκολη συζήτηση που θα την καταλήξει η διακυβερνητική ή το επόμενο κοινοβούλιο. Ποιες θα είναι δηλαδή οι σχέσεις της Ευρωζώνης με τις χώρες που αποφάσισαν να μην μπουν και να μην βάλουν χρήματα στο σχετικό ταμείο. Γιατί μπορεί και οι πολίτες και φορολογούμενοι των χωρών εκείνων να έχουν πρόβλημα από ό,τι αποφασιστεί. Καλή τύχη λοιπόν για τους επόμενους βουλευτές. Στους επόμενους βουλευτές. Μάλιστα, ο Βέρνερ σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ συμφωνώ ότι ε, κατά την επόμενη θητεία ίσως να χρειαστούμε πράγματι ένα νέο όργανο ελέγχου. Και όμως ε, που περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται, προβλέπονται μόνο ακροάσεις. Άρα δηλαδή μιλάμε για λάθος οργάνωση και έχει δίκιο η Σάρον. Στην αρχή είπε ότι δύο φορές απορρίψαμε και την τρίτη φορά έγινε μία πρόταση από τη γραμματεία και από ό,τι φαίνεται αυτή η πρόταση πέρασε από τους συντονιστέ σε αντίθεση με τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου το Προεδρείο επιθυμεί τώρα να αποφασίσει για μια υποεπιτροπή. Νομίζω ότι το θέμα για να συζητηθεί σωστά είναι τον Ιούλιο, στην επόμενη θητεία και όχι τώρα. Πρόεδρος, ε, πολλοί ε, θέλουν να λάβουν το λόγο. Διαδικαστικό θέλετε εσείς. Ναι, διαδικαστικό. Είναι πολύ λεπτό το θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν αποφασίσαμε και δεν είναι σημερινό θέμα. Γιατί ο κύριος Λάγκεν το άρχισε. Το βρίσκω άτοπο και παράκτερο. Εγώ αρνούμαι να πάρω θέση σε μια συνεδρίαση που δεν προέβλεπε αυτό το θέμα. Αλλιώ θα είχα και εγώ πολλά να πω προ τη θέση του Κοινοβουλίου έναντι του, της Ευρωζώνης, αλλά δεν είναι το δικό μας θέμα σήμερα αυτό. Όλε για το διαδικαστικό. Εγώ θα εξαρτηθώ από την απόφαση των συντονιστών και της Προέδρου. Επί της ουσίας, αν πάρετε μια τέτοια απόφαση για την επόμενη εντολή, δεν θα είναι κάτι τόσο φω γιατί θα διαιρέσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη και το Κοινοβούλιο. Μην το κάνετε αυτό αν θέλετε και άλλες χώρες να ενταχθούν στην Ευρωζώνη βέβαια. Κοιτάξτε πρέπει να κλείσει αυτή η συζήτηση. Θα το θέσουμε στην ημερήσια διάταξη σε κάποια φάση όταν θα έχουμε χρόνο. Jean Γκοζές, θα ήθελα ένα πράγμα να πω. Δεν είναι στην μερισία διάταξη, έχω ή έχει δίκιο, όλοι Αλλά θα πρέπει να αποδώσουμε τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Η κοινή επιστολή, την οποία συνυπογράψαμε, εκφράζει τις αποφάσεις τις οποίες κατέληξαν οι συντονιστές. Αυτό το οποίο δημιουργεί προβλήματα είναι αυτά που κάνουν στη διάσκεψη των Προέδρων και η γραμματεία του Κοινοβουλίου η οποία αντίθετα από ό,τι λέμε εμείς συνεχίζει να κρατάει τις δικές της απόψεις <clears throat> και καθορίζει με δύσκολο τρόπο το χρονοδιαγράμματα των συναντήσεών μας. Λοιπόν, τώρα δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τίποτα. Αν κάτι πρέπει να αλλάξει, αυτό θα το αποφασίσει το επόμενο κοινοβούλιο. Όπως είπε και η Σιλβή, ε, τα θέματα είναι κρεμή. Πρέπει να τελειώσουμε με αυτή τη συζήτηση τώρα και να την κάνουμε τη συζήτηση επί της ουσίας. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνει η συζήτηση λοιπόν τώρα. Ο Ζαν έκανε ένα σωστό σχόλιο. ότι υπήρξαν πιέσεις και από πλευράς του Γενικού Γραμματέα και γι' αυτό συζητάμε τώρα και γι' αυτό το θέμα αυτό ήταν στην επικαιρότητα ε, για αρκετό καιρό. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στη συζήτηση με τον Μπενουά Κιωρέ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο σημείο 13 της ημερησίας διάταξης, δραστηριότητες της Τρόικα. Thank you very much for being here uh, so punctually. Um, σας ευχαριστώ που ήρθατε στην ώρα σας. Okay, so Λοιπόν, λέει η Πρόεδρος. Προχωράμε λοιπόν ως ε, συνήθως, ε, δηλαδή καλωσορίζω τον ε, εισηγητή μας που έρχεται και πάλι στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε στην ακροασή μας και ελπίζω όταν θα έχουν σταματήσει οι συζητήσεις ε, θα μπορέσω να σας δώσω το λόγο για 10 περίπου λεπτά έτσι ώστε να παρουσιάσετε τις δικές σας σκέψεις και μετά ε, θα ε, προχωρήσουμε με τις ερωτεπαντήσεις. Μπενουά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα σας καθησυχάσω, θα τα πω αγγλικά. Ναι. Και εγώ και οι δύο συνεισηγητές και η Επιτροπή σας είχαν την ευγενή καλοσύνη να με καλέσουν. Η Τρόικα δημιουργήθηκε το 10 υπό ιδίως ιδιαίτερες συνθήκες, λειτουργήσε καλά κατ' εμάς. Θα επανέλθω σε λίγο. Αλλά βέβαια ε, πρέπει να πάρουμε και μερικά μαθήματα γιατί αναπτύσσεται η κρίση και ήδη οι χώρες βγαίνουν από τα προγράμματα. Οι δε μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν σε πολλές χώρες έχουν αρχίσει να καρποφορούν. Πρέπει λοιπόν συλλογικά να πάρουμε μαθήματα από ό,τι έγινε και να αρχίσουμε να αναλύουμε ποια θα μπορούσε να είναι μια μονιμότερη λύση για την κρίση στην Ευρωζώνη. Η συζήτηση εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί το Κοινοβούλιο προφανώς ως Ευρωπαϊκό Όργανο θα, θα, θα πρέπει να τα σκεφτεί αυτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκλησή σας. Είναι για μας πολύ σημαντικό. Περνάω τώρα στη γλώσσα του Σέξπιρ. Um, σας ευχαριστώ και στα αγγλικά για την πρόσκλησή σας για να καταλαβαίνουν και όσοι δεν ξέρουν. Ε, οι χώρες μέλη που αντιμετώπισαν την κρίση βρέθηκαν μπροστά σε μια πρόσμενη κατάσταση που επηρέασε τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών. Και γι' αυτό εσείς που είστε άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι θα έχετε κάνει την ανάλυση σας φαντάζομαι και είναι καθήκον νομίζω για όλα τα ευρωπαϊκά όργανα να πάρουν μαθήματα από ό,τι έχει γίνει και να βελτιώσουν τα πράγματα και η σημερινή συζήτηση είναι γι' αυτό πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εξηγήσω το ρόλο της ΕΚΤ στην Τρόικα αλλά και να παρουσιάσω την αξιολόγησή μας των προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν σε διάφορες χώρες και να πάρουμε και μερικά μαθήματα για το μέλλον. Αν μου το επιτρέπετε λοιπόν κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να πω μερικά λόγια για το ρόλο της ΕΚΤ στην Τρόικα που είναι και ο σκοπός της συζήτησής μας εδώ και δεύτερον να δούμε ποια είναι η αξιολόγηση που κάνουμε για τις διαδικασίες και τα μέτρα που ελήφθησαν και τρίτον να βάρουμε μερικά συμπεράσματα και μαθήματα για το μέλλον. Πρώτον λοιπόν να πω μερικά λόγια για το ρόλο της ΕΚΤ στην Τρόικα. Και θα κάνω τώρα, θα ανοίξω μία προσωπική παρένθεση. Δέκα μέρες μόνο εργάζομαι στη θέση που έχω και γι' αυτό ε, να με συγχωρήσετε αν δεν ξέρω τα πάντα για μυστικές συνομιλίες που μπορεί να έχουν γίνει σε διάφορους διαδρόμους της Ευρώπης γιατί δεν ήμουν παρόν. Αρχίζω υπενθυμίζοντας υπό ποιες συνθήκες δημιουργήθηκε η Τρόικα. Όταν ξέσπασε η κρίση την άνοιξη του 10 στην Ευρωζώνη, ακολουθούσε μία προηγούμενη βαρύτατη κρίση για την οποία δεν ήμασταν προετοιμασμένοι η αρχιτεκτονική του Μάστριχτ δεν είχε καταφέρει να εξισορροπήσει τα πράγματα και σε πολλές χώρες η Ευρώπη δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση ούτε υπήρχε κανένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση της έλλειψης πρόσβασης στις αγορές ορισμένων χωρών. Κανένα εργαλείο για χρηματοδότηση. Αυτή ήταν η κατάσταση την άνοιξη του 10. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση λοιπόν αποφασίσαν τα κράτη-μέλη να δώσουν, να χορηγήσουν χρηματοδοτική βοήθεια και προγράμματα διάσωσης με βάση ό,τι καλύτερο υπήρχε από τεχνογνωσία για τέτοια προβλήματα και τότε το Διεθνές Ταμείο και η Κομισιόν μαζί με την ΕΚΤ για να, για να συμπληρώνονται οι εμπειρίες τους και των τριών οργάνων για τη διαχείριση κρίσεων, η δημοσιονομική σταθερότητα κλπ. αποφάσισαν να αναδημιουργήσουν την Τρόικα. Τώρα ειδικά η έκτη τεχνογνωσία είχε εμείς στα δημοσιονομικά, στη μακροοικονομική σταθερότητα και ακόμα πιο σημαντικά ειδικά στην Ευρωζώνη, είχαμε τεχνογνωσία. Και γι' αυτό συμμετέσχαμε στην Τρόικα. Αλλά το ξεκαθαρίσαμε ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει την πλήρη της ανεξαρτησία, όπως προβλέπουν οι συνθήκες. Δεχόμενοι λοιπόν την πρόσκληση αυτή, δεχτήκαμε ότι θα έχουμε συμβουλευτικό ρόλο. Οι θεσμοί της Τρόικας δίνουν στην Ευρωζώνη τη δυνατότητα να λάβει αποφάσεις στο Eurogroup τουλάχιστον και εμείς αξιολογούμε εναλλακτικές δημοσιονομικές λύσεις και παρακολουθούμε, επιτηρούμε την εφαρμογή τους. Αυτή ήταν η απόφαση του Μαΐου 10. Σήμερα υπάρχει πια το ESM και στο δίμετρο του ΠΑΚ που εγκρίθηκε από κοινού με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Δεν αναφέρει βέβαια το ρόλο της ΕΚΤ. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφαση Sprinkle καθόρισε ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες της Ένωσης για τη συμμετοχή της ΕΚΤ στην Τρόικα μαζί με όσα προβλέπουν οι συνθήκες βέβαια. Να είμαστε λοιπόν σαφείς η συμμετοχή της ΕΚΤ στην Τρόικα έχει πολύ σοβαρή νομική υπόσταση. Δεύτερον, για τα προγράμματα προσαρμογής. Θέλω να τονίσω ότι παρά τις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων των διαφόρων χωρών, υπήρχαν και, κοινά, και κοινές προκλήσεις λανθασμένες εθνικές πολιτικές που δεν είχε αποτρέψει η πολιτική του Μάστριχτ φταίει και αυτό βέβαια όχι μόνο οι μεμονωμένες χώρες ήταν η βάση οι χώρες μέλη που είχαν προβλήματα δεν εφάρμοσαν πλήρως αυτά που προβλέπαν οι συνθήκες και πρόκειται λοιπόν και για συλλογική έλλειψη και φταίξιμα, πτέσμα. Σε κάθε μία από τις χώρες με πρόγραμμα η ΕΚΤ όπως είπε και ο πρώην πρόεδρος της Ζαν Κλοντ Τρισέ τον συναντήσατε και εσείς η ΕΚΤ είχε μιλήσει ήδη από πριν για απώλεια ανταγωνιστικότητας και υπερβολικούς μισθούς. Δεύτερον, Δεύτερη κοινή πρόκληση. Υπήρχε παρή μεγάλη πίεση χρόνου και οι πληροφορίες που υπήρχαν ήταν, δεν ήταν πλήρες και καμιά φορά και παραπλανητικές. Και αυτό κοινή πρόκληση σε όλες τις χώρες με πρόγραμμα. Τρίτον, οικονομικά, δημοσιονομικά προβλήματα αλλά και πολιτικά που καθιστούσαν την ευρωπαϊκή μέχρι τότε χρηματοδότηση ανεπαρκή και τέταρτον ελάχιστη εμπειρία για αντιμετώπιση κρίσεων μέσα σε συνθήκες νομισματικής ένωσης που μπορεί να δημιουργήσουν, να διαδώσουν την κρίση και σε άλλες χώρες. Όλα αυτά έπρεπε να ληφθούν υπόψη για να μην επεκταθεί η κρίση σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Αυτά ήταν τα κριτήρια με τα οποία λειτουργήσε η Τρόικα και οι συστάσεις της ε, ήταν κομμένες και ραμμένες στα προβλήματα της κάθε χώρας. Με στόχο απασχόληση και επαναφορά στις αγορές. Τρία θέματα χρειάστηκε να τονιστούν. Πρώτον, η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Δεύτερον, αναδιάρθρωση του νομισματικού και τραπεζικού τομέα και τρίτον ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και τα τρία έπρεπε να εφαρμοστούν ταυτόχρονα για να υπάρξει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και επαναφορά στις αγορές, επιστροφή στις αγορές. Θα ήθελα να τονίσω ότι όταν κάναμε συστάσεις ως τμήμα της Τρόικας, εμείς στην ΕΚΤ πάντοτε τονίζαμε την ανάγκη κοινωνικής δικαιοσύνης και αυτό σήμαινε η ισότιμη κατανομή των βαρών σε ολόκληρη την κοινωνία, σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Θα επανέλθω σε αυτό αν θέλετε αργότερα. Βεβαίως γνωρίζουμε πολύ καλά τις κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι χώρες με πρόγραμμα. Πολλές ακόμα τις υφίστανται. Γιατί έχασαν άνθρωποι τη δουλειά τους, μειώθηκαν οι μισθοί τους και οι συντάξει τους και αυτό μας ανησυχεί όλους. Αλλά να μην βγάλουμε το λάθος συμπέρασμα, ότι φταίει δηλαδή ο πυροσβέστης για τη φωτιά. Σκεφτείτε τι θα ήταν η εναλλακτική λύση. Οι χρεοκοπίες θα κατέστρεφαν τον, ε, δημοσιονομικό, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και αυτών των χωρών και άλλων. Και να μην ξεχνάμε ότι σε μία περίπτωση έγινε μεγάλη συζήτηση και για πιθανή έξοδο από την Ευρωζώνη. Τι έγινε λοιπόν τελικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τεράστιες προσπάθειες για την επαναλειτουργία, τη σωστή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα και εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Η Ιρλανδία, παραδείγματο χάρη, μόλι βγήκε από το πρόγραμμα και επέστρεψε στι αγορέ. Και αυτό δείχνει τι μεγάλη επιτυχία που είναι. Είδαμε ότι έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος και στον τομέα των δημοσιονομικών και σε σχέση κυρίως με τη σταθεροποίηση του πιστοτικού τομέα. Σταθερότητα των τιμών, αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και έχει βελτιωθεί επίσης και η πρόσβαση στις αγορές. Δυστυχώς η ανεργία παραμένει πολύ υψηλή, συνεπώς είναι έφραστη η ανάκαμψη και δεν θα πρέπει να αρκεστούν οι κυβερνήσεις στις προσπάθειες που έχουν γίνει. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τις χώρες σε πρόγραμμα, αλλά το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες παρατηρήσεις τελικές, ίσως συμπεράσματα, ίσως σε τρία επίπεδα. Πρώτον, τα προγράμματα ήταν η απαραίτητη απάντηση ε, σε χώρες οι οποίες ήταν ένα βήμα πριν από την πτώχευση. Δεύτερον, η Τρόικα ήταν στην συγκεκριμένη χρονική φάση το καλύτερο μέσο. Και τρίτον, λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες δυσκολίες και τις ατελείς πληροφορίες που είχαμε τότε, η Τρόικα μπόρεσε να δώσει σωστές συμβουλές. Πού βρισκόμαστε τώρα. Η εμπειρία των τελευταίων τεσσάρων χρόνων μας δίνει κάποια ενδιαφέροντα, θα έλεγα, μαθήματα. πάντα είναι κυρίαρχο να εμένει κανείς σε σωστές δημοσιονομικές πολιτικές έτσι ώστε οι χώρες αυτές να μην αντιμετωπίσουν εκ νέου μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία φυσικά και για τις νέες διαδικασίες εποπτείας, για το υπερβολικό έλλειμμα. Έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά θα ελεγχθούν στην εφαρμογή τους και σε καλές εποχές, όχι μόνο σήμερα. Αυτό είναι βασική ευθύνη φυσικά των ιδίων των κρατών μελών για να το πετύχουν. Γενικότερα είπαμε εμείς ότι η έλλειψη της σωστής διακυβέρνησης του πλαισίου αυτού σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο ευρωζώνης μείωσαν τις πολιτικές επιλογές που είχαμε. Μόνο όταν δημιουργήθηκε σταδιακά ένα νέο πλαίσιο άρχισαν κάποιες επιλογές να γίνονται διαθέσιμες και γι' αυτό εμείς ε, ε, καταλήξαμε στο ότι για να μπορέσουν να, να διατηρήσουν την οικονομική τους κυριαρχία τα κράτη-μέλη πρέπει να μοιραστούν εν μέρη αυτή την κυριαρχία. Είμαι βέβαιος ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσει να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο όπως μέχρι σήμερα. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι η Τρόικα στην παρούσα φάση δεν θα υπάρχει για πάντα Είμαι πεπισμένος ότι μακροπρόθεσμα το πλαίσιο διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενταχθεί σε μία ομπρέλα κοινοτικών νομικών ρυθμίσεων. Και εμείς θα συνεχίσουμε μαθαίνοντας από τις εμπειρίες να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ε, Πράγματι, με τον προκάτοχό σα ε, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι η Τρόικα δεν είναι τέλεια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε και κάτι άλλο καλύτερο αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά το ΕΛΚ, θα μιλήσει κάποιος από το ε, ΕΛΚ, Ότμαρ και επίση και συνηγητής, συνεισηγητής με συγχωρείτε, ε, της έκθεσης για την Τρόικα. Ότμαρ, έχετε το λόγο. Αξιότιμη κύριε Κορέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, εισήγησή σας ε, και πρέπει να πω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία είπατε. Όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα διότι στις επισκέψεις που είχαμε στα κράτη-μέλη αποκομίσαμε την εντύπωση ότι η Τρόικα δεν ε, έχει μόνο συμβουλευτικές ε, αρμοδιότητες και αρμοδιότητες ανάλυσης, αλλά μέσα στην ίδια την Τρόικα γίνεται μια πολύ έντονη συζήτηση σχετικά με την κατεύθυνση των προγραμμάτων. Και θα αναφερθώ σε δύο πράγματα που αναφέρατε. Ε, καταρχήν είπατε ότι ήταν μια έκτακτη κατάσταση, ότι δεν ήμασταν ε, προετοιμασμένοι για αυτήν και ότι η Τρόικα δεν θα υφίσταται εσαΐ. Και γι' αυτό λοιπόν ε, σας ερωτώ από την ε, εμπειρία σας ε, εντωμεταξύ μετά την Τρόικα ποιο είναι το όργανο εκείνο που θα ήταν ενδεδειγμένο και τι ακριβώς προτιμάτε εσείς για να σας βοηθήσει στην εκπλήρωση των καθηκόντων σας. Επίσης, στην αρχή είπατε ότι ε, δεν υπήρχε νομική βάση και μόνο με το του και με τη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης. Μόνο έτσι προέκυψε μία ε, βάση για τις δραστηριότητες ε, της Τρόικα. Και ερωτώ, αυτή η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η ύπαρξη της Τρόικας αρκεί και αυτή η θέσπιση βάσης άλλαξε τη δουλειά σας ή όχι. Δηλαδή, εξακολουθείτε να παραμένετε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και αν ε, ναι, τότε πώς ακριβώς επεκτάθηκαν οι αρμοδιότητές σας και σήμερα πώς ακριβώς θα διαμορφώνατε την δουλειά της Τρόικα και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όχι κάτι γενικό, γιατί γενικά μας είπατε. Κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί πολύ συγκεκριμένα πρέπει να πούμε στους πολίτες, όπως είπατε και εσείς, ότι αυτά που έγιναν έγιναν γιατί ήταν μια έκτατη κατάσταση, αλλά τώρα εργαζόμεθα για να υπάρχει μια μόνιμη βάσει ένα μόνιμο όργανο με βάση το κοινοτικό δίκαιο. Έτσι λοιπόν κατά την άποψη τι πήγε στραβά και τι ε, συμπεράσματα πρέπει να εξάγουμε από όλο αυτό το εγχείρημα. Okay, thank you very much, Mr. Uh, Ευχαριστώ κύριε συνεισηγητά. Θα σας απαντήσω με τη σειρά στα ερωτήματά σας. Πρώτον για το νομικό βάση, νομική βάση. Πράγματι, η συνθήκη του ESM και η Δήμετρος καθόρισαν τις ευθύνες της Κομισιόν και της ΕΚΤ μέσα στην Τρόικα. Ιδιαίτερα ως προς το ESM και το Διοικητικό του Συμβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε καμία βάση το 10 όταν άρχισε η Τρόικα. Η ΕΚΤ έχει ρόλο στήριξης γενικά των οικονομικών πολιτικών της Ένωσης με βάση βέβαια την ανεξαρτησία της και την εντολή της. Και τα προγράμματα προσαρμογής έπεφταν μέσα στην εντολή αυτή. Επίσης έχει το ρόλο η ΕΚΤ να επιτηρεί τη λειτουργία του νομισματικού συστήματος και δημοσιονομικού, δηλαδή χρηματοπιστωτικού συστήματος και το 125.5 το λέει αυτό. 127.5 με συγχωρείτε. Ο ρόλος μας λοιπόν στην Τρόικα ήταν εμπολής να στηρίζουμε την Ευρωζώνη για να διασφαλίζουμε οικονομική σταθερότητα. Και αυτό το λέει η συνθήκη. Υπάρχουν όμως και νέα όργανα όπως το ESM και η ιδρυτική του συνθήκη τα αποσαφήνισε ακόμα περαιτέρω. Επίσης, τα όργανα λήψης αποφάσεων του ESM, το διοικητικό του συμβούλιο δηλαδή στο Eurogroup, καθώς και του EFSM και EFSF έχουν καθοριστεί. Και το Δουνουτού βέβαια έχει δικά του όργανα λήψης αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δουνουτού. Οι αποφάσεις λοιπόν λαμβάνονται από αυτά τα σώματα και αυτό είναι και το σωστό. Γιατί πρόκειται για πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από σώματα υπόλογα σε πολιτικά όργανα. Επομένως και η ΕΚΤ και η Κομισιόν δεν μπορούν να αποφασίσουν μόνες τους. Και υπάρχει και ένας πρόσθετος λόγος γιατί η ΕΚΤ δεν μπορεί να αποφασίσει μέσα στην Τρόικα ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΤ πρέπει να διατηρήσει την πλήρη του ανεξαρτησία Όταν αποφασίζουμε λοιπόν για τη διάσωση ορισμένων τραπεζών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με πλήρη ανεξαρτησία, δεν δεσμεύεται από αποφάσεις είτε της Τρόικας είτε του ESM. Μετά λέτε ναι συζητήθηκαν τα προγράμματα στην Τρόικα. Βεβαίως συζητήθηκαν. Γι' αυτό και ήταν χρήσιμο. Και αυτό ήταν πολύ χρήσιμο γιατί αν δεν γίνονται συζητήσεις γιατί να έχουμε όργανα. Έχουμε τρία λοιπόν διαφορετικά όργανα που βλέπουν τα πράγματα με διαφορετικό πρίσμα. Το Δουνουτού πιο μακροπρόθεσμα, η Κομισιόν για να εκπληρώσει τον ηγετικό της ρόλο στην εποπτεία της λειτουργίας της Ένωσης και η ΕΚΤ έχει τη δική της οπτική γωνία, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη μακροοικονομική τη αυτή. Καμιά φορά διαφωνούσαμε. Αλλά μετά υπήρχε συμφωνία στην Τρόικα, αναφερόταν στην στο Eurogroup και το Eurogroup καμιά φορά έπαιρνε διαφορετικές αποφάσεις από τα συμπεράσματά μας. Αυτό το έχει πει και ο πρόεδρος Τρισέ. Η έκτα, που πούμε, αρχικά ήταν αντίθετη με το PSI στην Ελλάδα. Αλλά μετά αποφασίστηκε από το Eurogroup. Ήταν πολιτική απόφαση και θεμητή. Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μάλλον, με συγχωρείτε. Τώρα τα θέματα για το μέλλον. Τι θα αντικαταστήσει την Τρόικα. Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα της ΕΚΤ. Είναι θεσμικό θέμα. Δεν θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τι μόνιμο πλαίσιο θα υπάρξει. Ως κοινοτικό όργανο η ΕΚΤ φυσικά ενδιαφέρεται για την όλη διαχείριση των κρίσεων και για να υπαχθεί αυτή σε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο αλλά και για λόγους αποτελεσματικότητος πρέπει η πρόληψη και η διαχείριση των κρίσεων να συντονιστούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΕΚΤ δεν θα παίζει πια κανένα ρόλο. Παίζει ρόλο στη μακροοικονομική εξισορρόπηση όταν υπάρχει αποστολή σε κάποια χώρα. Είναι θέματα κοινοτικού νόμου, κοινοτικής νομοθεσίας. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι δεν θα παίξουμε κανένα ρόλο πια. Απλώς όλα αυτά θα υπαχθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Τον ίδιο ρόλο θα παίζει και τότε η ΕΚΤ. Πάντα θα υπάρχουν πολιτικές συζητήσεις και αποφάσεις δεν θα αποφασίζουμε εμείς. Ευχαριστώ. Ο άλλος συνεισηγητής, ο κύριος Γκόκ. Ευχαριστώ Σάρον. Καλημέρα Μπενουά. Σε ευχαριστώ για την παρουσίαση εδώ. Χαίρομαι που δέχθηκες αυτήν την συνάντηση. Δεν είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναδέχεται τέτοιες προσκλήσεις, πόσο μάλλον που ο ρόλος της εν πολύ συζητήθηκε και σχολιάστηκε και εννοώ ο ρόλος στο εσωτερικό της Τρόικα. Είναι καλό που είσαστε εδώ λοιπόν για να διευκρινίσετε τα πράγματα και ίσως να αρθούν και κάποιες ε, παρανοήσεις. Ξεκινώντας θα ήθελα να πω σε αυτά τα οποία ήδη σημείωσε ο Οτμαρ Το θέμα της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι σημαντικό για μας. Όταν δει κανείς το άρθρο 13 λέγεται ότι κάθε τέτοια συνταγματική ρύθμιση εντάσσεται στα πλαίσια ε, της συνθήκης. Εσείς λοιπόν πιστεύετε ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τράπεζας στο εσωτερικό της Τρόικα ανταποκρίνεται στην εντολή που της αποδίδουν οι συνθήκες. Ιδιαίτερα στα εξής θέματα, ίσως ένα αναθέμα στα οποία συζητήσαμε ήδη, για τα οποία συζητήσαμε ήδη. Να πω για την Ιρλανδία ότι εμείς συζητήσαμε με τον διοικητή της Κεντρικής Ιρλανδικής Τράπεζας. Και από ό,τι καταλάβαμε έγινε μια συζήτηση στο εσωτερικό της Τρόικα για το σχέδιο σωτηρίας των Ιρλανδικών πιστοτικών ιδρυμάτων. Η αίσθηση που δημιουργήθηκε είναι ότι κυριάρχησε στην Τρόικα η άποψή σας. Διαφορετική από τους άλλους, υπέρ ενός bail-out. Και ενώ η κυβέρνηση προτιμούσε ένα bail-in, το οποίο θα δημιουργούσε βέβαια θέματα στους ε, ε, μεγάλους κατόχους ομολόγων. Συμφωνείτε λοιπόν με την άποψη αυτή. Η απάντησή σας δεν είναι χωρίς συνέπειες γιατί ξέρετε ότι το bailout το πληρώθηκε από πολιτικές που επιβάρυναν τον Ιρλανδό φορολογούμενο. Και όταν λέτε ότι οι διαφορετικές πολιτικές ήταν απαραίτητες, να πούμε ότι η Ιρλανδία είναι διαφορετική περίπτωση. Γιατί έχει μια ευέλικτη αγορά εργασίας και τα δημοσιονομικά της ήταν σταθεροποιημένα πριν από την κρίση. Η αίσθηση στην Ιρλανδία σήμερα λοιπόν είναι ότι οι πολίτες πληρώνουν για μια κρίση για την οποία δεν φταίνε καθόλου. Και η Ιρλανδική κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να επιμικίνει την απόσβεση του χρέους της. Τα έχουμε συζητήσει και με τη Σάρων και θα ήθελα την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τι πιστεύετε γύρω από τις προτάσεις που έχουν γίνει από πλευράς Ιρλανδίας έτσι ώστε να βγει το τμήμα του Ιρλανδικού χρέους, το οποίο έχει σαν στόχο την σωτηρία των πιστοτικών ιδρυμάτων από τον υπολογισμό του ελλείμματος. Και τι πιστεύετε για κάποιες άλλες απόψεις για μεταφορά ενός τμήματος του χρέους του Ιρλανδικού στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, έτσι ώστε αναδρομικά να διαχειριστεί τη σωτηρία των τραπεζών. Για την Κύπρο θα είμαι πιο σύντομος. Υπήρξε μια απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας για να δοθεί μια ρευστότητα 9 δις στη Λαϊκή Τράπεζα η οποία παρόλα αυτά ε, ήταν γνωστό εκείνη την εποχή ότι δεν πήγαινε καθόλου καλά. Μπορείτε να δικαιολογήσετε την απόφασή σας και έρχομαι τώρα στα της Ελλάδας. Το καλύτερο για το τέλος. Συζητήσαμε επί μακρόν με τους εκπροσώπους του Δέλτα Νιτάφ και με τον κύριο Ρουμελιώτη συζητήσαμε στην Ελλάδα και από ό,τι φαίνεται είχαν υπάρξει σκληρές συζητήσεις ανάμεσα στο Δέλτα Νιτάφ και την Κεντρική Τράπεζα σχετικά με την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Το Δέλτα Νιτάφ μας είχε εξηγήσει ότι από την αρχή πίστευε ότι πρέπει να αναδιαρθρωθεί το χρέος γιατί πίστευε ότι δεν ήταν βιώσιμο και σήμερα είναι λιγότερο βιώσιμο γιατί ξεπερνά το 120% του ΑΕΠ που είναι ο, ο αριθμός το ανώτατο ποσοστό. Η στάση λοιπόν της Κεντρικής Τράπεζας τότε ήταν όχι στην αναδιάθρωση. Το Δέλτα Νιτάφ έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει αναδιάθρωση γιατί αλλιώς θα είναι πάρα πολύ βίαιη η δημοσιονομική εξυγίανση και θα δημιουργήσει προβλήματα στην ελληνική οικονομία. Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις στο Συμβούλιο τους επόμενους μήνες και τελικά υπήρξε η συγκεκριμένη γνωστή απόφαση. Λοιπόν, επιβεβαιώνεται ότι υπήρξε αυτή η συζήτηση στο εσωτερικό της Τρόικα. Επιβεβαιώνεται ότι σήμερα γίνεται μια νέα συζήτηση στο Συμβούλιο πλέον γύρω από μια νέα πιθανή αναδιάφραση του ελληνικού χρέους το οποίο θυμίζω ότι δεν θεωρείται βιώσιμο από το Δέλτα Νιτάφ. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, euh, δεν επιβαρύνθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης περίοδου. Αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλάβει ένα τμήμα των απολειών σε σχέση με αυτή την αναδιάρθρωση, αυτό θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε τις ζημίες αυτές να τις μόνο οι καταθέτες, οι τράπεζες και οι Έλληνες φορολογούμενοι. Ε, σας φαίνεται καλή αυτή η λύση γιατί έχετε θυμίζω 39 δις ε, στη διάθεσή σας ελληνικού χρέους. Ε, να σας ενημερώσω λιγάκι ότι έδωσα δυνατότητα στους δύο συνεισηγητές να κάνουν κατάχρηση χρόνου αλλά ε, δεν θα το επιτρέψω σε κανένα άλλον. Ο Ότμαρ ε, νομίζω ήταν δικαιολογημένο, αλλά μην ξεχνάτε ότι αν δεν έχουμε χρόνο τελικά οι άλλοι ομιλητέ ε, θα επιβαρυνθούν πολύ. Φαντάζομαι δηλαδή αυτό ισχύει και για μένα. Έχετε ήδη χάσει δύο λεπτά, λέει η πρόεδρος. Καταρχήν, ε, θα ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ότι χαίρεστε που η ΕΚΤ δέχτηκε την πρόσκληση. Δεν το καταλαβαίνω, έτσι και αλλιώς υποχρέωσή μας είναι να δεχόμαστε τις προσκλήσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και να πω επίσης ότι χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται ευκαιρία να λογοδοτήσω για το τι κάνει η Τρόικα. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει το σχετικό νομικό πλαίσιο, υπάρχει ε, και η διαδικασία των ερωταπαντήσεων και σε όποια ιδιαίτερη και έκτακτη ακρόαση οργανώστε, εμείς θα είμαστε παρόντες, δεν τίθεται καν θέμα επ' αυτού. Αυτά είναι θέματα αρχής για εμάς. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, κυρία Πρόεδρε, τέτοιαν πάρα πολλέ ερωτήσει και θα μπορούσα να μιλώ ώρε ολόκληρε για την κατάσταση στι χώρε αυτέ. Θα προσπαθήσω όμω να απαντήσω επί τη ουσία. Όσον αφορά την Ιρλανδία, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι η απόφαση να ε, προσφερθεί εγγύηση στι Ιρλανδικές Τράπεζε ελήφθη το 2008, δύο χρόνια πριν από την έναρξη του προγράμματο. Όταν άρχισε η εφαρμογή του προγράμματο ένα μεγάλο κομμάτι ε, του χρέους των ε, Ιρλανδικών τραπεζών είχε ήδη αποπληρωθεί. Δηλαδή ε, υπήρχε αυτή η απόφαση το, του Ιρλανδική, της κυβέρνησης πριν από την εμπλοκή της Τρόικας και αυτή ήταν μια διεθνή συμφωνία που είχε γίνει τότε, ότι δηλαδή οι συστημικές ε, τράπεζες έπρεπε να προστατεύονται από τις ε, κυβερνήσεις. Αυτό είπαν και οι G7 τον Οκτώβριο του 2008 έγινε στις ΗΠΑ, ε, στη Γαλλία, στη Γερμανία το είχαν όλοι αποδεχθεί αυτό, ότι οι συστημικές τράπεζες δεν θα έπρεπε να μπορούν να καταραίουν. Αυτή η απόφαση είχε ληφθεί κατά το παρελθόν. Έτσι λοιπόν αν τώρα τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αυτή η απόφαση πρέπει να αλλάξει όχι, νομίζω ότι έχει ήδη αλλάξει χάρη νημών. Δεν υπάρχει πλέον η EBRD ε, και από ό,τι φαίνεται κάποια στιγμή θα έχουμε έναν ενιαίο ε, μηχανισμό. Έχει προχωρήσει λιγάκι η όλη τοποθέτηση από το bailout στο bail-in. Πάντως ε, τότε η Διεθνή Συμφωνία ήταν να μην υπάρχει μετάδοση κρίσης από συστημικές ε, τράπεζες σε διεθνές επίπεδος και σίγουρα στην Ευρωζώνη. Τότε λοιπόν η ΕΚΤ ε, θεωρούσε ότι τα τραπεζικά δάνεια θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον κίνδυνο της συστημικής μετάδοσης. Έχουμε ξεφύγει τώρα από αυτό. Τότε όμως δεν είχαμε το σχετικό ε, νομικό πλαίσιο και κυρίως όσον αφορά την ε, Τράπεζα Ανασυγκρότησης ε, και Ανάπτυξης, την EBRD. Τώρα λοιπόν, επειδή παλαιότερα δεν είχαμε, τώρα έχουμε πλέον αυτό το πλαίσιο. Όσον αφορά τώρα την Κύπρο, η απάντηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίζει για ε, ενίσχυση ρευστότητας και αυτό μπορεί να εγκριθεί, να απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ε, ΕΚΤ. Τότε λοιπόν ε, υπήρχε η προοπτική ενός προγράμματος στήριξης που θα αφορούσε κυρίως την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Έτσι λοιπόν η, Εθνικός, Εθνική Υποπτική Αρχή, η Εθνική Τράπεζα δηλαδή της Κύπρου τότε ε, δούλευε βάσει της ε, παραδοχής ότι θα είχε κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό ε, πρέπει να υπάρχει ως προσέγγιση εφόσον ζητάει κανείς έκτακτη ενίσχυση ρευτότητας. Πρέπει να υπάρχει αυτή η δυναμική προσέγγιση. Η ειδική κατάσταση στην Κύπρο είναι ότι αυτό σύρθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί δεν προχωρούσαν οι συζητήσεις ανάμεσα στην τότε ε, κυβέρνηση της Κύπρου, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Τίμιο. Πάντως σας είπα, υπήρχε η παραδοχή ότι θα καταβάλλονται αυτά τα κονδύλια. Όταν όμως υπήρξε κίνδυνος να μην ε, υπάρξει αυτή η χορήγηση, τότε η Εθνική Τράπεζα της Κύπρου είπε ότι αν τελικά δεν καταβληθούν αυτά τα κονδύλια, τότε και δεν θα μπορούσε η τράπεζα να καταφύγει σε αυτό τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης. Ε, έπρεπε οπωσδήποτε να ε, δοθεί αυτή η έκτακτη υποστήριξη για να γίνει και πάλι, για να έχει η τράπεζα και πάλι ρευστότητα. Όσον αφορά τώρα στην Ελλάδα, πράγματι έγιναν συζητήσει για την αναδιάρθρωση του χρέου. Όμως το θέμα είναι ότι το PSI, το κούρεμα, θα μπορούσε παλαιότερα να προκαλέσει συστημική αναταραχή στην Ευρωζώνη. Αυτή ήταν η δική μας άποψη, αλλά και άποψη όλων των ευρωπαϊκών τραπεζών τότε, ότι τότε ε, δεν υπήρχε η δυνατότητα να ανταποκριθεί κανείς σε αυτή την ε, συστημική ευαισθησία. Και γι' αυτό το λόγο το 2010 δεν προβήκαμε σε περαιτέρω μέτρα γιατί αυτό θα είχε σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλες ε, τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Όσον αφορά ε, την τελευταία σας ερώτηση κατά πόν συζητείτε και πάλι αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, όχι δεν συζητείτε αυτό γιατί μέσα στην Ευρωζώνη και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουμε συμφωνήσει ότι η συζήτηση αυτή θα γίνει το 2014 σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους. Ε, η οι ε, συζητήσεις θα αφορούν το πρωτογενές πλεόνασμα ε, και την φορολογική πολιτική. Τώρα έχουν κατατεθεί κάποια στοιχεία τα οποία συζητούνται με την ελληνική κυβέρνηση. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ακόμα πιο σημαντικό, είναι ότι η Ελλάδα έχει προσαρμοστεί στο πρόγραμμα, καλύπτει τους στόχους της. Έτσι λοιπόν ελπίζουμε σύντομα να πάει η Τρόικα στην Αθήνα, να συζητηθούν περαιτέρω τα θέματα και κάποια στιγμή στα μέσα περίπου του 2014 θα επανέλθει η συζήτηση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς. Πρόεδρος, δεν έχουμε πια χρόνο που να μας ε, περισσεύει. Τα πέντε τα είχαμε εξοικονομήσει από προηγουμένως. Έτσι λοιπόν τώρα ε, θα έχουμε πάλι ε, περιορισμένο χρόνο. Γι' αυτό σας παρακαλώ θα ήθελα να είσαστε πιο ε, φιδωλή στις εκφράσεις Η Σιλβή. Ευχαριστώ. <coughs> Σάρων. Ακόμη και αν υπάρχει πίεση χρόνου θέλω να πω ότι κριμούμε ιδιαίτερα την παρουσία του κυρίου της ΕΚΤ γιατί όπως είπε και ο κύριος Γκοκ είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα και δείχνεται ότι είστε ανοιχτοί στο διάλογο. Έχω ένα ερώτημα πολύ συγκεκριμένο, απλό αλλά και ταυτόχρονα πολύπλοκο. Κάνουμε ό,τι πρέπει μακροπρόθεσμα δηλαδή. Συζητήσαμε για την ε, συγκυρία κτλ. αλλά στις χώρες των προγραμμάτων αρχίζει να, αρχίζουμε να έχουμε να διαφαίνεται κάποια προοπτική θετική. Διαρθρωτικά εννοώ διαρθρωτικά. Πολύ δύσκολο ερώτημα και δεν μπορώ να απαντήσω ναι ή όχι. Να με συγχωρεί η πρόεδρος. Μπορούμε να απαντήσουμε με δύο τρόπους. Πρώτον, ο καλύτερος τρόπος να προετοιμαστεί το μέλλον είναι να μεταρρυθμιστεί η οικονομία, να γίνει πιο ευέλικτη. Αυτό το λένε και τα προγράμματα. Και ισχύει και για το μέλλον, διότι έτσι η οικονομία γίνεται πιο ικανή να υποστεί δοκιμασίες. Και ιδιαίτερα να ανθίσει στις διεθνείς αγορές. Γι' αυτό χρειάζεται μια πιο ευέλικτη οικονομία παντού, όχι μόνο στις <coughs> αγορές των προγραμμάτων. Είναι η πρώτη απάντηση. Τώρα, αν το θέμα είναι αν έχουμε σαφή άποψη και όραμα για το πώς πρέπει να ειδικευτεί βιομηχανικά η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Κύπρος σε 10 ή 15 χρόνια, η απάντηση είναι όχι. Αν μου επιτρέπετε κάποιο σκεπτικισμό θα έπρεπε μάλλον να δαπανηθεί περισσότερος χρόνος για να βρεθεί τι ειδίκευση θα μπορούσε να έχει βιομηχανικά η κάθε χώρα στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας και μετά να σχεδιάσει εργαλεία εφαρμογής αυτής της πολιτικής αναδιάρθρωσης του εργατικού δυναμικού κτλ. Στην κρίση αυτή ένα από τα κύρια μαθήματα για μένα, το λέω προσωπικά, είναι ότι από τις μεγαλύτερες ελλείψεις που έχουμε στην Ευρώπη είναι ότι είναι ότι όταν συγκρίνουμε τη διαχείριση κρίσεων στην Ευρώπη και αλλού συνήθως καλούμε την Παγκόσμια Τράπεζα. Εμείς δεν έχουμε ανάλογα εργαλεία. Δεν μπορεί η ΕΤΕ να παίξει αυτόν τον ρόλο. Δεν θέλω να προτείνω τίποτε για την ΕΤΕ, έχει δική της εντολή. Παίζει σημαντικό ρόλο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πολλά μέρη της Ευρώπης αλλά εδώ εννοώ ότι τα εργαλεία υπάρχουν ίσως, αλλά δεν έχουν συνδεθεί με μια σφαιρικότερη στρατηγική. Ευχαριστούμε ο Φίλιππος. Ευχαριστούμε κύριε Κερέ. Δύο ερωτήσεις και μπορείτε να απαντήσετε με ναι ή όχι. Φανταστείτε σε μια υποθετική περίπτωση ένας ισπουνός πρωθυπουργός να στείλει μια απόρριτη επιστολή στην ΕΚΤ και παραπονιέται για την νομισματική πολιτική η οποία βλάπτει τα συμφέροντα της χώρας του και αυτό είναι αλήθεια βέβαια το επόμενο, μια επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στον Πρωθυπουργό τον Ισπανό λέγοντάς του ότι πρέπει να κάνει αλλαγές στην αγορά εργασίας. Απλή ερώτηση. Πιστεύετε ότι η πρώτη περίπτωση είναι αποδεκτή και η δεύτερη περίπτωση και αυτή, αν είναι αποδεκτή ή όχι. Τρίτο θέμα, και μπορείτε να μου απαντήσετε και γαλλικά, θα κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Λοιπόν, τον Μάιο του 10 είχατε πει ότι είστε κατά της αναδιάφασης του ελληνικού χρέους, γιατί αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό το που ο Λίαμ μας είπε για την Ιρλανδία δεν είναι αναχρονιστικό, γιατί ήδη το 11 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απειλεί την Ιρλανδική κυβέρνηση να διακόψει τη βοήθεια προς τα πιστοτικά ιδρύματα της χώρας αν η κυβέρνησή της δεν πληρώνει αυτά τα οποία δεν εγγυήθηκε. Δηλαδή να καλύψει την πιθανή απώλεια των μεγάλων καταθετών. Λοιπόν, και απαντήσατε τότε σε αυτούς που διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν θέλετε να υπάρξει απειλή στη δημοσιονομική σταθερότητα και οι δύο αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προστατεύουν τους ιδιώτες ε, καταθέτες αντίθετα ε, με ε, το ευρύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Για να το πω λίγο πιο απότομα, δεν είναι ορθολογικές οι απόψεις αυτές και δεν δείχνετε να έχετε εμπιστοσύνη στις αγορές. Ταυτόχρονα όταν υπάρχει απειλή επιμόλυνσης αν θέλετε, αυτό σημαίνει διότι ε, ένα μεγάλο ποσοστό του δημοσίου χρέους κρίνεται μερικές φορές μη επιστρέψιμο. Συγγνώμη πρόεδρε καθυστερώ αλλά είναι σημαντικά αυτά τα θέματα μπορούμε να διατηρήσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα με διαφορετικό χώρο, κάνοντας αναδιάρθρωση του ιδιωτικού και του δημοσίου χρέους όταν αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να επιστραφεί το χρέος αυτό, ότι δεν είναι βιώσιμο. Εσείς λοιπόν ποιον προασπίζεστε σήμερα, μήπως αντί να προασπίζεστε την κοινωνία, προασπίζεστε τα ιδιωτικά πιστοτικά συμφέροντα. Hang Χωρίς μικρόφωνο. Δεν θα ανεχθώ τέτοιου είδου στάση. Πήρατε πάρα πολύ χρόνο από τον διαθέσιμο. Παρακαλώ απαντήστε. Ευχαριστώ. Να πω ότι το ότι συζητάω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι μια κοινωνική ενασχόληση, είναι υποχρέωση. Ναι και ναι στις πρώτες ερωτήσεις σας. Αν θέλει η Πρόεδρος μπορώ να σχολιάσω. Οι κυβερνήσει ασκούν πάντα κριτική στη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, Ένα ε, υπουργό οικονομικό μεγάλη χώρα τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι το, η αξία του ευρώ είναι πάρα πολύ υψηλή και αυτό δημιουργεί προβλήματα κτλ. Κριτική μα ασκείται συνεχώ. Σε όλε τι χώρε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει συμβουλέ στις κυβερνήσεις και οι κυβερνήσει λαμβάνουν υπόψη τι συμβουλέ ή όχι, πολύ συχνά όχι. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε σύμβουλοι των κυβερνήσεων σε θέματα οικονομικά απλά. Ναι και ναι στις πρώτες ερωτήσεις σας λοιπόν για την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εμείς είπαμε ότι το πέρασμα από τον κόσμο του bailout στον κόσμο του bail-in είναι θετικό. Υποστηρίξαμε εμείς την οδηγία για τις πιστωτικές κρίσεις. Θα θέλαμε να πάμε ακόμα περισσότερο προς κάποιες κατευθύνσεις, αλλά απαιτείται για να γίνει αυτό ένα πλαίσιο. Και εκείνη την εποχή, πριν δύο-τρία χρόνια, δεν είχαμε την οδηγία, δεν υπήρχε γενικότερη συζήτηση για το Μπέιλιν ούτε στο Συμβούλιο Οικονομικής Σταθερότητας και δεν υπήρχε αν θέλετε firewall, δεν υπήρχε προφυλακτήρας που θα επέτρεπε να γίνει πιο ανθεκτική η Ευρωζώνη. Αυτό έγινε με τον μηχανισμό σταθερότητας σε εύθετο χρόνο. Λοιπόν, αυτά για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Τώρα που υπάρχουν οι νέοι κανόνες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ισχυρότερη, η έννοια της λογοδοσίας έχει τονιστεί ακόμα περισσότερο και τα λάθη πληρώνονται. Ευχαριστώ. Είστε τυχερός που μπορείτε να μιλάτε και στα γαλλικά. Ο Γιούργεν Κλούτε για την ΚΟΕ. Εγώ μιλάω όμως γερμανικά. Δεν ξέρω γαλλικά και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Κύριε Κορέ, σας ε, καλωσορίζω θερμά. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε. Ε, θα είμαι ως το δυνατόν πιο σύντομος γίνεται. Η αποστολή της ΕΚΤ είναι σε νομισματική πολιτική, σταθερότητα, πολιτική χρήματος. Είπατε ότι η ΕΚΤ είναι σε θεσμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως ως τέτοιος δεσμεύεστε από τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα κοινωνικά δικαιώματα στο οποίο είναι προσιλωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ορίζεται και σε πάρα πολλές αποφάσεις ε, δικαστηρίων. Επ' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ερωτώ λοιπόν, αυτή ε, τη σχέση με τα κοινωνικά δεδομένα. Τι λαμβάνετε υπόψη σας σε όλα αυτά τα οποία αποφασίζετε. Γιατί ξέρετε, σε τελική ανάλυση οι αποφάσεις σας έχουν κοινωνικές συνέπειες και αυτό το είπατε και εσείς στην εισαγωγική σας παρέμβαση. Ε, Έτσι λοιπόν, η δέσμευση της ε, ΕΚΤ, η προσήλωσή της στα θεμελιώδη δικαιώματα και τα κοινωνικά δικαιώματα δεν θα έπρεπε να οδηγήσει η ΕΚΤ ε, να λάβει υπόψη της τις κοινωνικές συνέπειες, άρα δηλαδή κατόπιν τούτου να λάβει άλλου είδους μέτρα. Και πίσω από όλα αυτά ε, υπάρχει το εξής ερώτημα σε μια τέτοια έκτακτη περίπτωση που πραγματικά δεν μπορούσε να προβλεφτεί, ε, που δεν ήμασταν έτοιμοι, σωστά όλα αυτά, αλλά μπορεί κανείς τα κοινωνικά δικαιώματα να τα ε, παραβιάσει και σε μεγάλο βαθμό και να τα καταργήσει αν θέλετε με τέτοιο βάναψο τρόπο. Αυτά που σας είπα έπαιξαν ρόλο στις αποφάσεις τις οποίες έλαβε η ΕΚΤ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά εγώ πρέπει να φύγω και η κυρία Λούλινγκ έχει την καλοσύνη να αναλάβει το συντονισμό της συζήτησης. Και ζητώ συγγνώμη. Κοιτάξτε και αυτή είναι μια σημαντική ερώτηση. Αναμφίβολα η ΕΚΤ δεσμεύεται από το κοινωτικό πλαίσιο και από τις ε, διεθνείς ε, συμφωνίες. Όλα αυτά αφορούν βέβαια ανθρώπινα δικαιώματα και που δεν είδα θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι η ΕΚΤ δεν δεσμεύεται από αυτές τις συμφωνίες. Προφανώς και δεσμεύεται. Να ξεκαθαρίσω όμως ένα πράγμα, ότι η προσαρμογή ήταν απαραίτητη. Ήταν λοιπόν απαραίτητη απαραίτητο να βρεθούν νέε ισορροπίες ε, στις οικονομίες, ε, να υπάρξει κάποια ευθυγράμμιση ε, των δαπανών και γενικότερα της απόδοσης αυτών των οικονομιών. Νέες λοιπόν ισορροπίες, άρα δηλαδή νέα προσαρμογή. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το επιτύχει κανείς αυτό. Αυτό που εμείς προσπαθήσαμε και εξακολουθούμε να προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι κάτι το οποίο να είναι κοινωνικά δίκαιο, δηλαδή το βάρος της ε, προσαρμογής να μην επιβαρύνει υπέρμετρα τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα και χαμηλότερα εισοδήματα. Ε, σίγουρα έχει τους νέους και τους ε, ηλικιωμένους. Αυτό είναι θέμα δικαιοσύνης και μετά υπάρχει και το θέμα της αποτελεσματικότητας, δηλαδή να γίνει τέτοια προσαρμογή που να είναι και αποτελεσματική. Και θα αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα για να γίνω κατανοητός. Ήταν απαραίτητο να περιστούν σε όλες αυτές τις χώρες οι δημόσιες δαπάνες, γιατί δεν ήταν πλέον βιώσιμες και γιατί οι κυβερνήσεις ε, χρηματοδοτούσαν αυτές τις δαπάνες με ξένα χρήματα. Άρα δηλαδή ε, δεν ήταν δικά τους τα χρήματα για την χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών. Βεβαίως η προσπάθεια της προσαρμογής έπρεπε να γίνει με έναν τρόπο ανάλογα με το επίπεδο εισοδημάτων. Είπαμε στην ΕΚΤ, η ΕΚΤ στην Ελλάδα, η περικοπή των ε, συντάξεων και των μισθών θα ήταν ανάλογα με το ύψος αυτών, άρα δηλαδή διαφοροποίηση. Κατόπιν είπαμε ότι έπρεπε να βελτιωθεί η ίσπραξη φόρων να υπάρχουν περισσότερες ε, φορολογικές ε, κλίμακες για να γίνεται καλύτερη κατανομή στην κοινωνία. Αυτό αποδείχτηκε πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο να γίνει η αλλαγή, αλλά και αυτό θεωρούσαμε ότι είναι ε, στοιχείο δικαιοσύνης. Και ένα τρίτο στοιχείο αφορά τον ανταγωνισμό τον τομέα των προϊόντων και της παραγωγικότητας. Σε αυτές τις χώρες βλέπουμε πραγματική αλλαγή στο μοναδιαίο κόστος εργασίας. Ε, διαπιστώσαμε πράγματι ότι υπήρξαν ε, πολλές απολύσεις. Αλλαγή λοιπόν του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Και πρόσφατα βιώσαμε και προσαρμογή των τιμών. γιατί τι νόημα έχει η μείωση του μοναδιαίου κόστου εργασίας και καμία προσαρμογή των τιμών. Αυτό απλά σημαίνει ότι ε, το βάρος το φέρουν μόνο τα νοικοκυριά. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει και προσαρμογή της ε, τιμής ε, των προϊόντων να υπάρχει καλύτερος ανταγωνισμός, αυτό να ισχύει στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και αλλού, έτσι ώστε η προσαρμογή να κατανεμηθεί δικαιότερα και να μην φέρουν το σύνολο του βάρους μόνο τα νοικοκυριά. Ε, νομίζω αυτά είναι σημαντικά. Ο κύριος Γκοζές. Κοιτάξτε κύριε κύριε, σας ευχαριστώ, αλλά αφήνω το λόγο στον κύριο Φεγιό. Έτσι θα έχει λίγο περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ. Θα αρχίσω, θα αρχίσω λέγω, συγχαίροντάς σας για αυτά που μόλις μας είπατε. και που γεννούν στο μυαλό μου τρία ερωτήματα. Πρώτον, μπορείτε να μας πείτε τίποτε περισσότερο για το τι θα είχε γίνει στις τέσσερις αυτές χώρες αν δεν είχαν εφαρμοστεί αυτές οι έκτακτες λύσεις της Τρόικας. Τι θα είχε γίνει. αν δεν είχε βρεθεί αυτή η λύση για τις χώρες που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Μπορείτε να μου το απαντήσετε και με οικονομικούς όρους αλλά και με κοινωνικούς γιατί συμφωνώ ότι ήταν πολύ σημαντική κοινωνική πτυχή. Τι εξέλιξη θα είχε σημειωθεί στον κοινωνικό τομέα αν οι λύσεις της Τρόικας δεν είχαν εφαρμοστεί. Δεύτερον, νομίζετε ότι υπήρχαν πραγματικοί κίνδυνοι για το σύνολο της Ευρωζώνης. Δηλαδή, υπήρχε πραγματικός κίνδυνος εξόδου χωρών από την Ευρωζώνη και τι επιπτώσεις θα είχε αυτό για το σύνολο της ζώνης. Τέλος, τρίτον δηλαδή, εγώ είμαι Πορτογάλος και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την παρούσα κατάσταση των τεσσάρων αυτών χωρών στα προγράμματα. Η μία βγήκε από αυτά, η Πορτογαλία ετοιμάζεται να τελειώσει σε τέσσερις μήνες. Υπάρχουν θετικοί και ενδείξει για την οικονομία της, αλλά μπορείτε να μας πείτε τίποτε παραπάνω. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Φεγιό για την ερώτησή του τι θα είχε συμβεί χωρίς τη στήριξη της Ένωσης και του Δέλτα Νιτάφ. Μιλάμε για χώρες που είχαν χάσει την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, που δεν μπορούσαν να, να χρηματοδοτήσουν τις υποχρεώσεις τους. Θα είχαν πτωχεύσει ουσιαστικά. Οι τράπεζες είχαν επενδύσει σε δημόσιο χρέος και αυτό θα οδηγούσε στην καταστροφή του χρηματοπιστωτικού τομέα, πτωχεύσεις, ο κόσμος θα έτρεχε να αποσύρει τα χρήματά του, οι καταθέτες θα χάναν τα χρήματά τους, γιατί προστατεύονται μέχρι τις 100.000, αλλά παρόλα αυτά όταν το ίδιο το κράτος έχει ουσιαστικά πτωχεύσει τότε δεν θα βοηθήσει κάτι τέτοιο. Η εξωτερική βοήθεια ήταν απαραίτητη. Και η εξωτερική βοήθεια βοηθάει και την κατανομή του κόστους και της προσπάθειας προσαρμογής σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και η ευρωπαϊκή βοήθεια και η βοήθεια του Νιτάφ επέτρεψαν να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες του χρέους, υπερβολικές δημόσιες δαπάνες, υπερεπέμβηση σε ορισμένους τομείς, σε ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα στις κατοικίες. Βοήθησε τις χώρες και τις ε, κυβερνήσεις των χωρών να κάνουν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και όχι σε σύντομο χρονικό διάστημα με την πίεση των κεφαλαίων αγορών για να το πω σε πολιτικό επίπεδο. Η προσπάθεια αυτή βοήθειας βοήθησε τις χώρες αυτές να ελέγχουν πάντα τη διαδικασία προσαρμογής. Πολύ δύσκολη η διαδικασία βέβαια και είναι πάντα δύσκολη. Αλλά η εξωτερική βοήθεια κατέστησε ικανές τις χώρες αυτές σε συνεργασία με την Ένωση και το ΔΕΛΤΑ να σχεδιάσουν την προσαρμογή με ελεγχόμενο τρόπο γιατί αλλιώς αυτό θα είχε γίνει μέσα σε λίγες ημέρες και λίγες εβδομάδες με άτακτο τρόπο, με πολύ μεγάλη σύγχυση και δεν θα έλεγχαν τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν uh, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον υπήρχε κίνδυνος γενικότερα στην Ευρωζώνη. Πράγματι υπήρχε κίνδυνος λόγω της αλληλένδεσης ε, και της ε, έκθεση σε ομόλογα ε, σε διάφορες χώρες της Ευρωζώνης. Άρα δηλαδή υπήρχε ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης, υπήρχε ο κίνδυνος η κρίση να μεταφορθεί και σε άλλες χώρες της ε, Ευρωζώνης. Τέλος, ε, η ερώτηση σχετικά με το ποια είναι η κατάσταση σήμερα, ας πούμε στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο στην εφαρμογή του προγράμματος. Ε, το πρόγραμμα εκτελείται ε, όπως ε, προβλεπόταν. Αυξάνεται το ΑΕΠ, έχουμε ανάπτυξη. Η ανάπτυξη οικονομίας έχει μειωθεί η ανεργία, άρα δηλαδή οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Νομίζω αυτό θα το αποφασίσει η κυβέρνηση της ε, Πορτογαλίας γιατί όπως είπατε ε, μέσα σε λίγους μήνες ε, θα ληφθεί η απόφαση ή θα αποφασιστεί κατά πόσον η Πορτογαλία σιγά σιγά θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα ή κατά πόσον θα ακολουθήσει ένα δεύτερο πρόγραμμα. Πάντως επαναλαμβάνω για την Πορτογαλία η πρόοδο της είναι εντυπωσιακή. Ο κύριος Μπούλμαν έχει το λόγο. Κύριε Κορέ, πρέπει να πω εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά που μας λέτε. Η τοποθέτησή σας είναι πολύ συμπαθητική, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα δεδομένα και τα στοιχεία. Γιατί βλέποντας τα στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, διαπιστώνω ότι το δημόσιο χρέος και η ανεργία αυξήθηκαν δραματικά. Ε, στην Ελλάδα, α πούμε, η ανεργία έχει σχεδόν διπλασιαστεί, αλλά και στην Πορτογαλία. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Γι' αυτό λοιπόν πολύ με ενδιαφέρει να μάθω. Η ΕΚΤ που είναι αρμόδια για την νομισματική πολιτική, μα η νομισματική πολιτική καθίσταται όλο και πιο δύσκολη σε μια ευρωζώνη όπου οι ισχυροί γίνονται ισχυρότεροι και οι αδύναμοι πιο αδύναμοι. Πώς μπορείτε λοιπόν, λοιπόν να βρείτε μια ισορροπία με αυτές τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Από τη μια έχουμε την ΕΚΤ η οποία συνάπτει μνημόνιο συναντήληψης ε, και με βάση αυτή την συμφωνία καθίσταται η νομισματική πολιτική ακόμα δυσκολότερη την οποία καλείται να αντιμετωπίσει με άλλες συμφωνίε. Αυτό είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι εξή σχετικά με τι επενδύσει. Εμείς προτείνουμε τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. 11 χώρες θέλουν να εισάγουν αυτό το φόρο, αλλά εσείς εμφανίζεστε ε, στην κοινή γνώμη όλο και πιο απρόθυμοι και η κοινή γνώμη ε, έχουν την εντύπωση ότι τα χρηματοψηφιακά Ινστιτούτα εκβιάζουν, εκβιάζουν ε, κυρίαρχα κράτη να μην εφαρμόσουν αυτό το φόρο. Εσείς όμως, ξέρετε, εκπροσωπείτε την τραπεζική εποπτεία και θέλω να μας πείτε το επιβεβαιώνεται αυτό ότι ασκείται τρομακτική πίεση όχι μόνο στη Γαλλία, προφανώς στη Γαλλία, αλλά και στην Ιταλία και στη Γερμανία. Κοιτάξτε, όσον αφορά τη δική μου την πατρίδα, τη Γερμανία, ξέρω πάρα πολύ καλά πως οι ενώσει τραπεζών ε, προσπαθούν να αποτρέψουν κυρίαρχα κράτη, όπως σας είπα, να εισάγουν αυτό το φόρο. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως μια εποπτική αρχή ε, που στηρίζει ποτέ την Ευρωζώνη, πώς ακριβώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό. Έχετε ακόμα δυόμιση λεπτά για να απαντήσετε. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω μέσα σε αυτό το χρόνο. Λοιπόν, αυτά που είπατε για την ανεργία ή την απασχόληση στην Ελλάδα και την Πορτοκαλία είναι σωστά. Όταν λέμε ότι βελτιώνονται τα πράγματα, μιλάω για τα τελευταία στοιχεία που έχουμε. Τους τελευταίους μήνες του 2013 δηλαδή. Φυσικά η ανεργία αυξήθηκε πάρα πολύ μεταξύ 10 και 13 φυσικά. Ιδιαίτερα η ανεργία των νέων όπως είπατε κι εσείς. Έχει παραπάνω από διπλασιαστεί. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι είναι μια αναπόφευκτη διαδικασία σε μια κρίση να γίνουν οι προσαρμογές και στις άλλες χώρες βέβαια, σε ολόκληρη την Ευρωζώνη αλλά ακόμη περισσότερο στις χώρες των προγραμμάτων. Η ανεργία αυξήθηκε, οι χρεοκοπίες αυξήθηκαν κλπ. ως αποτέλεσμα των μέτρων. Αυτό που είπα είναι ότι σιγά σιγά βλέπουμε θετικά στοιχεία όπως αυξημένη ανταγωνιστικότητα και άρα περισσότερες εξαγωγές. Οι εξαγωγές είναι μέρος της ζήτησης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι προσπάθειες αυτές σιγά σιγά αποφέρουν καρπούς. Αλλά συμφωνώ απόλυτα ότι είναι μόνο τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν κάτι θετικό ως βελτίωση στις οικονομίες αυτές. Πιστεύω όμως ότι τα σημεία είναι αληθινά, ιδιαίτερα ανταγωνιστικότητα, εξαγωγές και για την Πορτογαλία ίσως και ανεργία. Τώρα αν η ΕΚΤ συμβάλλει στην κατανομή των βαρών στην Ευρωζώνη λόγω κρίσης, εγώ πιστεύω ότι τα προγράμματα που εφαρμόζονται συμβάλλουν στη σύγκληση. Άρα καταπολεμούν τον κατακαιρματισμό που φοβάστε. Ας πούμε η ανταγωνιστικότητα πάλι. Μπορούν οι χώρες έτσι να ολοκληρωθούν περισσότερο μέσα στην ενιαία αγορά. Είναι και αυτό μια σύγκληση. Γιατί οι εξαγωγές καταρχήν πηγαίνουν προς άλλες χώρες της Ένωσης. Βλέπουμε πολύ μεγάλη σύγκληση και στα πιστοτικά. Κυβερνήσεις όπως και πρόσφατα στην Πορτογαλία μπόρεσαν να ξαναμπούν στην αγορά και να εκδώσουν ομόλογα. Αυτά είναι σύγκληση και σιγά σιγά έτσι θα διευκολυνθεί η δουλειά της ΕΚΤ που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ από τον κατακαιρματισμό που αναφέρατε. Τέλος το FTT, μία φράση για το FTT, για το FTT. Αυτό είναι ε, φορολογική πολιτική, δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Συμφωνούμε, αλλά το FTT λέμε ότι πρέπει να στοχεύει έτσι ώστε να μην εμποδίζει τα υπόλοιπα προγράμματα. Εμείς δεν έχουμε τίποτε κατά του FTT. Ναι, είναι νέα αντίληψη αυτή, γιατί ο κύριος Ντράγκη και ο κύριος Τρισέ ήταν πάντα αντίθετοι. Αλλά Ούντο, ε, νομίζω ότι πήρες μια πάρα πολύ καλή απάντηση και δεν πρέπει να εστιάζεσαι. Κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, χαριτωμένοι είσαστε ε, όπως ε, πάντα. Εδώ όμως μιλάμε για σοβαρά θέματα και ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτά που μας είπε. Κυρία Κράτσα, κυρία Κράτσα έχετε το λόγο. αυτό που θέλω να σας ρωτήσω κύριε Κιωρέ, είναι σε συνέχεια αυτό, αυτό που ήδη ανέφεραν συνάδελφοί μου, οι κοινωνικές επιπτώσεις της κατάστασης αυτής και από τη μεριά την ηθική, από τη μεριά του σεβασμού του κοινοτικού κεκτημένου, αλλά και από τη μεριά των στοιχείων της ανάκαμψης. Στην Ελλάδα αυτό το μεγάλο ποσοστό ανεργίας, κυρίως των νέων ανθρώπων και η φυγή των νέων εκπαιδευμένων ανθρώπων είναι ανασταλτικά για την ανάκαμψη η οποία πρέπει πάση θυσία να έλθει. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είπατε ότι ο πυροσβέστης δεν φταίει, εννοώντας την Τρόικα, τα προγράμματα προσαρμογής, ε, δεν έχει κάνει απολογισμό ο πυροσβέστης. Τα, οι λάθος πολλαπλασιαστές που έχουν αναφερθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η έλλειψη κατάλληλων σταθεροποιητών για την ε, κοινωνική συνοχή και το ρόλο της στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάκαμψη αυτά δεν έχουν υπολογιστεί μήπως στην περίοδο αυτή που η Τρόικα κάνει την τελευταία της αξιολόγηση στην Ελλάδα πρέπει να γίνει μια από εσά σύσταση αλλά μας αποδείξατε ότι είναι πολιτικές οι αποφάσεις που παίρνονται αλλά από εσά μια εμφανή σύσταση ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα αυτά για να δοθεί αυτή η ανάσα που χρειάζεται και η ελληνική κοινωνία αλλά και η ελληνική οικονομία για να έχει ένα νόημα αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο επετεύχθη με τεράστιες θυσίες και σταθερή προσέγγιση, θυσίες από το λαό και σταθερή προσέγγιση από την κυβέρνηση. Διότι και στη φορολογία δεν έγιναν μόνο οι κατάλληλες προσαρμογές που έπρεπε να γίνουν, οι κατάλληλες μεταρρυθμίσεις, έγινε υπερφορολόγηση. Η οποία υπερφορολόγηση βαρύνει και την αναπτυξιακή διαδικασία και την κατανάλωση. Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο που είμαστε, εσείς που είπατε ότι δίνετε σημασία σε αυτό το τομέα, για την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανάπτυξη, νομίζω ότι θα έπρεπε να το δείτε σε αυτό το πλαίσιο. Θα είναι πολύ σημαντικό η συστάση σας και για τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρθουν στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ για το ερώτημα. Για τους πολλαπλασιαστές δεν θα μακρηγορήσω. Φυσικά οι πολλαπλασιαστές το 10 ήταν υψηλότεροι, αποδείχτηκαν υψηλότεροι από ό,τι αναμέναμε. Αλλά δεν είναι επιστήμη εδώ η οικονομετρία. Ό,τι και να πούμε για τα αποτελέσματα της εξυγίανσης επηρεάζονται από πάρα πολλούς παράγοντες όπως και την αξιοπιστία μεταξύ άλλων των πολιτικών των προγραμμάτων δηλαδή για να μειωθεί η δυσπιστία των αγορών που ήταν μεγάλο πρόβλημα για αυτές τις χώρες δεν είχαν πρόσβαση στις αγορές. Είναι ένα απλό παράδειγμα. Λοιπόν, είναι πιθανό ο πολλαπλασιαστής ούτως ή άλλως να είναι όπως τον αναγνώρισε το Δουνουτού. Υπάρχει μια διαδικασία εκμάθησης εδώ πειραματισμού. Τώρα για το περιεχόμενο των προσαρμογών, φόροι και δαπάνες. το σύνολο της ΕΚΤ και άλλων οργάνων της Τρόικας υπενθύμησαν στις εθνικές κυβερνήσεις τα δυσάρεστα αριθμητικά στοιχεία. Δηλαδή αν δεν έχετε πρόσβαση στις αγορές και χρειάζεστε χρηματοδότηση, τότε πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή είτε προς τις δαπάνες είτε προς το αντίθετο. Από τους φόρους δηλαδή. Αυτό είναι απλή αριθμητική. Φυσικά η φύση των περικοπών των δαπανών μπορεί να συζητηθεί και να συζητηθεί και το είδος της φορολόγησης. Η φορολόγηση φυσικά πρέπει να είναι προοδευτική, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε είτε την περικοπή των δημοσίων δαπανών είτε την αύξηση των φόρων. Γιατί δεν έχουμε πια εξωτερική χρηματοδότηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λεωνάρδος Δομήνικη. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξή. Διάβασα κάποιες ε, πρόσφατες ε, παρεμβάσεις και πρέπει να πω ότι μου άρεσαν ιδιαίτερα γιατί βρήκα σε αυτές ε, κάποια πολιτική και πολιτιστική ευαισθησία που δεν συναντά κανείς συνήθως σε άτομα που έχουν αξίωμα όπως το δικό σας. Εσείς μας είπατε ότι η κρίση είναι μια διαδικασία από την οποία μαθαίνει κανείς, βγάζει συμπεράσματα και νομίζω μιλήσατε και για την αξιολόγηση της διαδικασίας προσαρμογής. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δεν πιστεύετε κι εσείς ότι το πρόβλημα είναι περισσότερο ο τρόπος, η μορφή με την οποία εκτελέστηκαν αυτά τα προγράμματα προσαρμογής. Γιατί δεν αναφέρομαι τόσο στην κατάσταση σε συγκεκριμένες μεμονωμένες χώρες, αλλά αναφέρομαι περισσότερο στο ότι δεν υπήρχε ε, κάποιο σύστημα που να εφαρμοστεί και που να διέπει αυτές τις διαδικασίες προσαρμογής. Δηλαδή, ε, οι διαδικασίες αυτές ε, θα μπορούσαν να έχουν κάποια επιτυχία μόνο εάν εκλαμβάνει κανείς την Ευρωζώνη ως μια ζώνη ενιαία για να επέλθει ισορροπία. Εσείς όμως λέτε ότι είναι θέμα πολιτικό και είναι και θέμα νομικής φύσεως. Όμως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ό,τι λέει είναι πολύ σημαντικό. Άρα δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί κατά κάποιον τρόπο να πει στους πολιτικούς τι είδους μαθήματα πρέπει να εξάγουν. Και με αυτό θέλω να τελειώσω. Κατά τη δική μου άποψη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει στα χέρια της μια πολύ σημαντική ε, δικλίδα ασφαλείας, δηλαδή τον πληθωρισμό του γύρω 2%. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο και θα μπορούσε κανείς επίσης να σκεφτεί ότι ε, και η αύξηση των τιμών στις πιο ισχυρέ χώρες, αυτό επίσης θα μπορούσε να είναι ένα κομμάτι μιας πολιτικής επαναφοράς της ισορροπίας. Τρία λεπτά έχετε στη διάθεσή σας για να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Βουλευτά. Και τώρα πάλι στη γλώσσα του Σέξπιρ. Συμφωνώ ότι φυσικά παίζει ένα ρόλο η ΕΚΤ για να προειδοποιεί τις κυβερνήσεις ότι υπάρχει κίνδυνος στη λειτουργία της Ευρωζώνης ή για την ακαιρεότητά της. Και το είδαμε αυτό μέχρι και το 12. Τώρα πια δεν υπάρχει νομίζω τέτοιος κίνδυνος. Και κατά πόσον βέβαια υπάρχουν, να προειδοποιεί αν υπάρχουν κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών. Γι' αυτό ήμασταν χρήσιμοι στην Τρόικα να έχουμε αυτήν τη συστημική προσέγγιση στη διαχείριση των κρίσεων και είπαμε στις κυβερνήσεις από νωρίς ότι χρειάζονται firewalls. Τους είπαμε ότι χρειάζεται ένα συνοπτικό πλαίσιο για τις πτωχεύσεις τραπεζών. Δεν λέμε ότι όλα εμείς τα κάναμε, αλλά προειδοποιήσαμε ιδιαίτερα με τα Μπέιλιν. Και τώρα λέμε στις κυβερνήσεις ότι χρειάζεται ένας ενιαίος μηχανισμός επιλύσεων και εξυγίανσης και ταμείο. Και αυτό δεν πρέπει να καθυστερήσει πολύ αν θέλουμε να παίξει σταθεροποιητικό ρόλο για την Ευρωζώνη. Τα ξέρετε αυτά λοιπόν. Τέτοια μηνύματα δίναμε στις κυβερνήσεις. Μπορείτε να υπολογίζετε σε εμά ότι θα προειδοποιούμε πάντοτε όταν διακυβεύεται το συμφέρον της Ευρωζώνης στο σύνολό της. Το 2% του πληθωρισμού. Ε, είμαστε αποφασισμένοι να επιμείνουμε στον ορισμό μας τη σταθερότητα των τιμών, 2% δηλαδή μεσοπρόθεσμα. Και αυτό είναι απαραίτητο για να συνεχίσουμε να δίνουμε τις συμβουλές που δίνουμε. Αν δούμε, διαδούμε κανέναν κίνδυνο για την μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών θα αντιδράσουμε αμέσω. Ευχαριστούμε πολύ. Εξετίμησα ιδιαιτέρως αυτά που είπατε για το Ταμείο Εξυγίανσης. Λυπούμε που οι Γερμανοί του ΕΛΚ δεν είναι πια εδώ. Έχω ακόμη τρεις στον κατάλογο, κυρία Γκόμες, κύριο Σμιτ και Σβέν Γκίγκολντ. Επειδή έχουμε χρόνο, μπορούμε να τους ακούσουμε έναν έναν. Είχαμε πει καταρχήν όλους μαζί να απαντήσετε, αλλά μπορείτε και έναν έναν. Η κυρία Γκόμες πρώτο. Κύριε Κορέμου, η Τρόικα δεν έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων και στη συλλογή των φόρων. Γιατί η ΕΚΤ και η Τρόικα γενικότερα δεν το έκανε. Στην Πορτογαλία αυξήθηκαν πάρα πολύ οι φόροι της μεσαίας τάξης και των πτωχών, γιατί όμως δόθηκαν ε, φορολογικές ελαφρύνσεις σε εταιρείε που καταφεύγουν σε φορολογικούς παραδείσους. Γιατί χορηγήθηκαν φορολογικές αμνηστίες που δίνουν ασυλία στους μεγαλύτερους φοροδιαφεύγοντες και φοροφυγάδες που πληρώνουν μόνον 5,5% φόρο, 7,5% φόρο με συγχωρείτε. Ο κύριος Αλμπουκέρκε μας είπε όταν είχε έρθει ότι η διάσκεψη της Ντοβίλ τον Οκτώβριο του 10 όπου παρίστατο και ο Σαρκοζή και η Μέρκελ που μίλησε για τον ιδιωτικό τομέα δημιούργησε τελικά την κλιμάκωση των, της κερδοσκοπίας κατά του ευρώ. Δεν νομίζετε ότι και αυτό οδήγησε την Πορτογαλία μεταξύ άλλων να ζητήσει bailout. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Για τις λεπτομέρειες σχετικά με τα φορολογικά, όπως σας είπα, εμείς είμαστε ενός σταδιακού προοδευτικού συστήματος οι αποφάσεις τις οποίες αναφερθήκατε είναι αποφάσεις της πορτογαλικής κυβέρνησης. Και έρχομαι σε αυτά που λέγαμε πριν. Η Τρόικα δίνει συμβουλές, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις και έτσι πρέπει, γιατί αυτές είναι πολιτικά υπόλογες. Είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση δηλαδή γι' αυτό, για την Ντοβίλα. Γενικά η συζήτηση για το PSI είχε γίνει εκεί. Ξέρετε ότι εμείς δεν ήμασταν υπέρ και αυτό είχε πράγματι συνεισφέρει στην κλιμάκωση της κρίσης και στα προβλήματα του δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη. Δεν είναι ο μοναδικός λόγος βέβαια και αυτό χτύπησε κυρίως τις χώρες οι οποίες είχαν διαφθρωτικές ανισότητες, ναι. ανισορροπίες και η Πορτογαλία ήταν μια τέτοια χώρα και πράγματι αυτό προκάλεσε ε, την κλιμάκωση της κρίσης από εκεί και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Κιωρέ. Είπατε να μην κατηγορούμε τον πυροσβέστη για την πυρκαγιά. Ε, εσείς είσαστε από το 12 στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πιστεύετε ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες πρέπει να, να κατηγορηθούν γιατί δεν προειδοποίησαν για την κρίση. Γιατί για μένα αυτή η συνάντηση αφορά την ευθύνη και το υπόλογο του καθενός. Το θέμα δεν είναι τι κάνατε από εκεί και πέρα, αλλά νομίζω ότι έχετε κάποιες ευθύνες και για το γεγονός της κρίσης, για το ΔΝΤ υπάρχει μια συζήτηση για την πιθανότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού Δέλτα Είναι καλό κάτι τέτοιο ή μήπω χρειαζόμαστε την εμπειρία. Και τέλος για τα FTTs. Εγώ έρχομαι από τη Σουηδία, έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο φορολογίας και ήταν καταστροφική οι ε, προκάτοχοί σας είπαν ότι είναι μια κακή λύση και ένας κακός φόρος αυτός ο φόρος στις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Έχετε αλλάξει την άποψή σας <clears throat> γι' αυτό. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω σύντομα με το τελευταίο το φόρο των χρηματοψηφιστικών συναλλαγών, το FTT. Ε, μετά θα επανέλθω με περισσότερες λεπτομέρειε αν θέλετε. Κοιτάξτε, οποιαδήποτε φορολογία συμπεριλαμβανομένου και του φόρου αυτού είναι σωστή ανάλογα με τις ε, συνθήκε, ε, και καλό είναι να μην υπάρξουν μη προβλεπόμενε αντιδράσει, κυρίω όσον αφορά τι βραχυπρόθεσμε αγορέ. Εσείς προέρχεστε από τη Σουηδία, εγώ από τη Γαλλία όπου υπάρχει ένας τέτοιος φόρος, περιορισμένος βέβαια και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Δεν λέω απαραίτητα ότι αυτό είναι το σωστό πρότυπο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για να εφαρμόζεται ένας φόρος επί των χρηματοψηφιστικών συναλλαγών, ανάλογα με το πώς είναι σχεδιασμένος. Τώρα, κατά πόσον οι κεντρικοί τραπεζίτες θα έπρεπε να έχουν προειδοποιήσει νωρίτερα, ε, σας είπα, ε, πράγματι υπάρχει κάποια συλλογική ευθύνη όσον αφορά τη μη εφαρμογή ενός ε, πλαισίου. Τότε εγώ δεν ήμουνα ε, στην ΕΚΤ, αναφέρομαι περισσότερο στους προκατόχους μου. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ πριν από την κρίση, το 5, το 6 ως Ευρωζώνη είχε προειδοποιήσει ότι η εξέλιξη των μισθών ήταν πάρα πολύ ψηλή, πάρα πολύ δυναμική σε αρκετές χώρες και κυρίως είχαν αναφερθεί ε, στο, στην ψαλίδα ανάμεσα στο μοναδίο κόστος εργασίας ε, ε, και τους δημόσιους μισθούς γενικότερα στην Ευρωζώνη. Ήταν σαφής από αυτού και νομίζω η ΕΚΤ είχε τοποθετηθεί όταν εξετάστηκε το 2003 το Σύμφωνο Σταθερότητας κυρίως όταν παραβιάστηκε αυτό από τις μεγάλες χώρες και υπήρχαν κάποια μηνύματα τότε στην εφαρμογή ε, του συμφώνου κάποια μηνύματα τα οποία είχε προβάλλει και επισημάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σχετικά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το ξεχάσατε αυτό. Κοιτάξτε, ως προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτή τη συζήτηση την κάνουν τα κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη, όπως ξέρετε, είναι μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχουν δηλαδή δικαίωμα να απευθυνθούν στο δούνου του, αν συμφωνήσει βέβαια και το δούνου του. Ε, όπως σας είπα, εγώ τάσομαι αναμφίβολα υπέρ του να επανέλθουν όλα κάτω από την ομπρέλα του κοινοτικού δικαίου. Και επίσης θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει κάποια συνέπεια. Το EIP, MIP, κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν αυτά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πια το δουνουτού. του. Αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν έχω συγκεκριμένη άποψη και αυτό που μπορώ να σας πω από το παρελθόν ήταν ότι η ε, συμμετοχή του Διεθνούς ε, Νομισματικού Ταμείου ήταν χρήσιμη γιατί έχουν εμπειρία, εμπειρία κρίσεων, ε, εμπειρία που δεν είχαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δούνο του λοιπόν ήταν το μόνο σκέλος στην Τρόικα που είχε αυτή την εμπειρία ε, χωρών ε, στα πρόθυρα της ε, χρεοκοπίας. Και νομίζω ότι είχαν πραγματικά μια αξιόλογη συμμετοχή. Να πω σε σχέση με αυτά τα οποία λέγατε προηγουμένως ότι πάντα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας προειδοποιούσε στη χώρα μου σαν παράδειγμα την προσαρμογή στον προπολογισμό των αμοιβών. Περνάμε στον τελευταίο ομιλητή, τον Σφεν Γκίγκολντ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι η οξύτητα κριτική κριτικής απέναντι σε κάποιες πράξεις της ΕΚΤ για μένα είναι μη δικαιολογημένη γιατί με τον τρόπο αυτό αυτό απλά τιμωρούμε εκείνον που αναλαμβάνει κάποια ευθύνη, να αντιμετωπίσει κάποια κατάσταση. Εσείς το κάνατε αυτό και αυτό ήταν σωστό. Ε, Δηλαδή εσείς αναλάβατε αυτό που δεν έκαναν τα κράτη-μέλη, που δεν ανέλαβαν τις ευθύνε τους και κατόπιν τούτου ε, ακούτε κριτικές ε, που όμως δεν έχουν καμία σχέση με την εντολή που σας έχει δοθεί και γι' αυτό είστε αναγκασμένος να ακούτε τέτοιου είδους πράγματα. Οι συστάσεις ε, τις ε, οποίες στηρίξατε μετά από έρευνες που έχουν γίνει αφορούν σε παραβίαση του ε, κάρτη του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και εσείς ε, τις ε, συστάσεις σας τις αιτιολογήσατε λέγοντας ότι μα αν δεν τα κάναμε όλα αυτά τότε η κατάσταση σε κοινωνικό επίπεδο θα ήταν ακόμα χειρότερη. Όμως, ξέρετε, όταν παραβιάζονται ε, θεμελιώδη δικαιώματα, αυτό δεν μπορεί κανείς να το προβάλλει σε επιχείρημα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιέρετα και αναλωτρίατα. Έτσι λοιπόν θέλω να σας πω ότι η θέση που πήρατε στην Τρόικα θεωρείται ότι αποτελούσε παραβίαση ανθρωπίων δικαιωμάτων, δηλαδή ενός ε, δικαίου το οποίο δεσμεύει και εσάς. Και το δεύτερο ερώτημά μου αφορά αυτό που είπε ο Γάλλος ε, συνάδελφος σχετικά με τη διάσωση της Λαϊκής ε, Τράπεζας στην Κύπρο με βάση τα προγράμματα έκτακτης ανάγκης είπατε ότι ε, χορηγήσετε βοήθεια σε αυτή την τράπεζα διότι θεωρήσατε ότι θα υπάρξει ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας. Όμως οι κανόνες για την ΕΚΤ απαγορεύουν κάτι τέτοιο. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι η ΕΚΤ μπορεί να βοηθήσει με την προσδοκία και την παραδοχή ότι θα υπάρξει ανακεφαλαιοποίηση. Γι' αυτό ρωτώ συγκεκριμένα, παραδέχεστε ότι παραβιάσατε το καταστατικό και κατόπιν τούτου και εσείς ε, κατά κάποιον τρόπο συμβάλλατε στο να βάλουν πόδι σε αυτή την τράπεζα οι ιδιώτες. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον ε, αφορά, μάλλον καταρχήν το πω αλλιώς, ε, σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή που κάνατε. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι για μας ο ρόλος της ΕΚΤ δεν είναι σε περίοδους κρίση ότι είμαστε μέλος μιας τρόικας. Εμείς ε, ανθρωπιστικά θέλουμε να συμβάλλουμε. Εντάξει, δεν θα το κουβεντιάσουμε σήμερα αυτό, αλλά εν πάση τόσο, ο δικός μας ο ρόλος ήταν να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα τιμών μέσα από ανθρωπιστική πολιτική και όπως ξέρετε το έχουμε κάνει αυτό με διάφορους τρόπους και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αυτό δεν συζητιέται σήμερα, για τα πρακτικά το λέω, αλλά αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χορηγεί συμβουλές στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης, ε, δεν λαμβάνουμε εμεί αποφάσεις. Αυτό έχει γίνει απόλυτα σαφές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν είμαστε τμήμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Απλά δίνουμε συμβουλές και τις αποφάσεις τις λαμβάνουν οι εθνικές κυβερνήσεις μέσα στο κοινοτικό πλαίσιο και η Ευρωζώνη. Όμως, διακόπτει ο μιλητής, αυτά που συμβουλεύσατε ήταν συμβατά με το διεθνές και το ευρωπαϊκό κοινωνικό δίκαιο. Γιατί αυτό Λέτε οι συνθήκε που σα δεσμεύουν. Και ρωτώ, εσείς δεν θεωρείτε ότι παραβιάσατε το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία σας. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι δικηγόρος, μην με στριμώχνετε με νομικής φύσεως θέματα. Εγώ θέλω να σας πω ότι η ΕΚΤ προφανώς και δεσμεύεται από τον νόμο και οι συστάσεις της Τρόικας αναφέρονται και δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λοιπόν μπορείτε και εσείς να ανατρέξετε και να ελέγξετε το τι ακριβώς συνέβη. Προφανώς και μας δεσμεύει το κοινοτικό δικαίωμα. Δεν θεωρούμε ότι είμαστε εκτός ε, κοινοτικού δικαίου. Να είναι σαφές αυτό. Όσον αφορά τον έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότησης, τον ELA αυτός ε, προβλέπεται στην περίπτωση της ΕΚΤ, αλλά εξαρτάται από την αξιολόγηση που θα γίνει για την φερεγγιότητα της τράπεζας. Τότε λοιπόν και ακόμα και σήμερα η αξιολόγηση αυτή γίνεται από αρμόδιες ε, εθνικές αρχές, άρα δηλαδή τότε στην Κύπρο την αξιολόγηση την έκανε η Εθνική Τράπεζα της Κύπρου. Και αυτό έγινε το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΚΤ πρέπει να βασίζεται σε μια αξιολόγηση την οποία την κάνει μια εθνική αρχή. Η ΕΚΤ δεν είχε και μέχρι τον Νοέμβρη δεν θα έχει εποπτικές αρμοδιότητες. Έτσι λοιπόν αυτός ο μηχανισμός ε, ε, προσφέρεται σε μια εθνική τράπεζα και τον κίνδυνο τον αναλαμβάνει η εθνική τράπεζα. Άρα δηλαδή εμείς είμαστε αναγκασμένοι να βασιστούμε σε αυτό που μας είπε η Εθνική Τράπεζα της Κύπρου. Η αξιολόγηση της ε, Εθνικής Τράπεζα Κύπρου και αυτό κοινοποιήθηκε ήταν ότι η λαϊκή ήταν φερέγγια υπό την παραδοχή ότι θα μπορούσε να καταφύγει σε αυτό τον μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης. Εμείς δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε γιατί σας είπα αυτή ήταν μια αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας της Κύπρου. Όταν όμως η ΕΚΤ θα έχει εποπτικές αρμοδιότητες τότε βέβαια θα αλλάξουν τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το μόνο που θέλω είναι να σε ευχαριστήσω για τις εξηγήσεις σας που συνέβαλαν σε μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και διάλυση παρεξηγήσεων. Ίσως να διορθώθηκαν έτσι και ορισμένες απόψεις προκαθορισμένες, προκατηλημένες. Ευχαριστώ όλους όσους έλαβαν το λόγο. Η επόμενη συνεδρία θα γίνει τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου στις 15 η ώρα. Τσακ τσακ.